Uh, ladies and Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να καθίσουμε. Έχουμε καθυστερήσει ένα τέταρτο. Περιμένω και τον συμπρόεδρο, τον Γκέι Μίτσελ. Από ό,τι όμως με ενημέρωσαν, έρχεται. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Σήμερα έχουμε μία κρόση για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Ανάπτυξης για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τόσο σημαντικό που το ξεχάσαμε. Και επειδή ακριβώς το, το ξεχάσαμε, ε, πρέπει τώρα να το θυμηθούμε και να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μια καταπάτηση όλων των Καταπάτηση λοιπόν ενός δικαιώματος των δικαιωμάτων ε, της γης αυτό δηλαδή που επέτρεψε στη Δύση να αναπτυχθεί Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν ήρθαν εδώ πλούσιοι άνθρωποι και έδωσαν ένα 0,7 ε, ε του ΑΕΠ τους ε, στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ και με αυτόν τον τρόπο κατέστησαν ευημερούσε οι χώρε αυτές. Στην ουσία, αν δούμε την ιστορία της ανάπτυξης, την κλασική ιστορία, η κλασική ιστορία είναι μια ιστορία όπου μια, ένα, ε, μια γη στην οποία δεν έμενε κανεί, ίσω έμεναν ορισμένε φυλέ, όπου δεν υπήρχαν ούτε δρόμοι, ούτε αυτοκίνητα, ούτε σχολεία, ε, ηλεκτρισμό, δεν υπήρχε τίποτα τέλο πάντων σε αυτή την γη. Ε, και μέσα σε 100 χρόνια αυτή η άγωνη γη έγινε ε, από τα πλουσιότερα μέρη του κόσμου. Αυτή είναι η ιστορία των Πολιτειών της Αμερικής. Δεν ήταν άνθρωποι με διδακτορικά από το Oxford ε, και το Cambridge, αλλά ήταν πρόσφυγες από την Ευρώπη. Αυτοί που πήγαν εκεί. Ήταν άνθρωποι που έφτασαν εκεί με τίποτα στα χέρια τους. μόνο με, με πολύ λίγα ρούχα, με ένα κουρέλι ε, ντυμένοι με ένα κουρέλι, οι οποίοι όμως ήταν έτοιμοι να δουλέψουν. Ήθελαν λοιπόν να εργαστούν σκληρά για να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Δεν θα μπορούσαν όμω να τα έχουν κάνει όλα αυτά, εάν δεν είχαν μια νομική δομή που να τους έδινε τη δυνατότητα αυτή τη σκληρή εργασία να τη μετατρέψουν σε κεφάλαιο, κεφάλαιο σε πλούτο, το, το πλούτο ε, σε επενδυτικά κεφάλαια και τελικά να φτάσουμε στο σύγχρονο καπιταλισμό. Και όλα αυτά μας δείχνουν ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε τίποτα ως δεδομένο. Στις Βρυξέλλες Κάποια στιγμή όλοι αγοράζουμε το σπίτι μας, ε, αγοράζουμε τη γη μας, την οποία θέλουμε συνέχεια να την ε, αφήσουμε στα παιδιά μας. Όλα αυτά τα θεωρούμε δεδομένα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αγοράζουμε μετοχές που είναι χαρτιά, αλλά που είναι τιτλοποιήσιμα αυτά τα χαρτιά και δημιουργούν πλούτο ή και δεν δημιουργούν όπως μας έδειξε η πρόσφατη ιστορία. all this is αλλά... taken όλα αυτά είναι μέσα, είναι εργαλεία που και πήραν αυτούς τους ε, ε, και ε, οι Ευρωπαίοι αυτοί που φορούσαν κουρέλια, που φορούσαν προδιές όπως σας είπα, έφτασαν εκεί και τελικά δημιούργησαν πλούτο. Ο πλούτος κατέστη δυνατός χάρη στη νομική αυτή δομή, με την οποία ε, υπήρξαν, τα, ε, ε υπήρξαν τίτλοι ιδιοκτησία, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Τώρα, ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά αλλού. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πληρώνουμε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ των φορολογούμενων στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως στην Αφρική για παράδειγμα, και όμως δεν αλλάζει τίποτα σαν αφορά αυτό το ζήτημα. Δεν αλλάζει τίποτα γιατί δεν υπάρχουν οι δομές για τη σώρευση κεφαλαίου, για τη σώρευση πλούτου. Που συνέχεια θα, τον θα, θα αφήσει τον πλούτο αυτό και στα παιδιά του. Και οι χώρε που έχουν αυτέ τι δομέ διέφυγαν τις φτώχεια. Οι χώρε που δεν έχουν αυτή τη δομή ε, είναι ε, κολλημένες σε αυτό το δικό τους σύστημα. Εάν αγνοήσουμε αυτό το γεγονός, ό,τι αναπτυξιακή βοήθεια και αν δίνουμε, ό,τι και να κάνουμε, χάνουμε το χρόνο μας. Το, το θέμα είναι το εξή. Πώ η Ευρώπη και η Αμερική ε, ε, έγιναν ε, ευημερούσε περιοχέ. Α, είναι απλό. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα το απόγευμα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι μιλώ και, και κερδίζω χρόνο και περιμένω να έρθει και στην πρόεδρο. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μια παμπάλαια έννοια στη χώρα μου, στην Βρετανία, ε, είχαμε διάφορα συστήματα μίσθωσης γης, ιδιοκτησίας μικρών ε, εργοστασίων, ε, μικρών εκμεταλλεύσεων, που, μικρών επιχειρήσεων που είχαν το δικαίωμα να τις πουλήσουν, είχαν, και τε, είχαν τεμάχια, αγροτεμάχια στα οποία φύλαγαν τις αγελάδες τους, τελικά πλήρωναν φόρο. Όλα αυτά τα θεωρούμε σαν δεδομένα, επαναλαμβάνω. Αλλά αν δούμε όμως αναπτυσσόμενες χώρες, παραγνωρίζουμε τελείω το γεγονό ότι δεν έχουν αυτά τα θεμέλια οι χώρε αυτέ. Πρόκειται λοιπόν για μια άσκηση ε, με την οποία θα σκάψουμε τα θεμέλια. Είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει σοβαρά το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν άλλοι σε άλλα σημεία της γης, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται εδώ, σε, αυτή την πλατφόρμα, έχουν αναλάβει το καθήκον αυτό και εργάζονται προ την κατεύθυνση αυτή. Πάντω, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε σοβαρότητα και από το πρίσμα, υπό το πρίσμα τη ανάπτυξη. Θα έχουμε δύο πάνελ σήμερα. Το πρώτο πάνελ θα εξετάσει τη σημασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησία και τη ίδια ιδιοκτησία ω βασικέ προκλήσει για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ε, στον τομέα τη γη σε αναπτυσσόμενε ε, ε, χώρε. Θα συζητήσουμε συγκεκριμένα εργαλεία και θα εξετάσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα επιτόπου. Ιδιαίτερα από τη Ρουάντα και τη Μαδαγασκάρη. Επίσης, έχω εδώ στο Προεδρείο ως μέλος του πάνελ τον Κλέιτον Σέφερ. Ο πατέρας του, Πίτερ Σέφερ, ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της χαρτογράφησης, ε, κτηματολογίου ε, και ε, οριοθέτησης εντοπισμού των δικαιωμάτων στη ΣΥΠΑ. Εργάστηκε με τον Πίτερ, με τον Τεσότο, φημισμένος οικονομολόγος που έγραψε πολύ σημαντικά βιβλία για το, πάνω στο γιατί γιατί ε, έγινε ο καπιταλισμός, ε, γιατί υπάρχουν ορισμένε φτωχέ και ορισμένε πλούσιε χώρε ε, και πώ θα ανέβουν την κλίμακα τη ιδιοκτησία σε διάφορε χώρε. Να και ο συμπρόεδρο, σε παρακαλώ, έλα στο Προεδρείο, σου κρατάω τη θέση. Και στα πλαίσια αυτά των έργων του Ντεσότο, που και του έργου του Ντεσότο, που το συνέχισε ο Πίτερ Σέφερ, έχουμε τώρα τον Κλέιτον, ο οποίος προσπαθεί να τα δει τα πράγματα από πιο πρακτική σκοπιά, χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Ο Κλέιτον Σέφερ, λοιπόν, ε, είναι επικεφαλής ε, στις ΗΠΑ Πολιτείες ενός ομίλου ε, Global Land Group Από πανεπιστημίου ε, στη ΣΥΠΑ και στην ε, Αβάνα. Νομίζω ότι ακολούθησε τα χνάρια του Μπάρακ Ομπάμα. Κλέιτον, σε παρακαλώ χωρίς να καθυστερώ άλλο, ε, πάρε το λόγο και πες μας την άποψή σου. Πες μας τι κάνεις, γιατί το κάνεις και τι προτείνεις. Σας ευχαριστώ. θέλω να μιλήσω για τα βαθιά θεμέλια της οικονομίας της αγοράς και πώς δημιουργήθηκαν. Ε, οι χώρε δωρητέ έχουν δαπανίσει πολλά χρήματα στα προγράμματα ε, για τα δικαιώματα ιδιοκτησία στο τελευταίο ήμιση του αιώνα, αλλά δεν έχουν δώσει τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Αυτοί που υποστηρίζουν τα δικαιώματα ε, ιδιοκτησία, όπω ο Ερνάντο Δεσότο, μα υποσχέθηκαν ένα είδο μετασχηματισμού των αναπτυσσόμενων χωρών. Τελικά όμω δεν έγινε αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε. Ω μέρο τη εργασία μου στα πλαίσια ε, του Global End Group, που είναι μια εταιρεία ε, συμβούλων και τεχνολογία ε, και εστιάζει την προσοχή τη σε χαρτογράφηση κτηματολογίου χαμηλού κόστου και σε ασφαλή μικροχρηματοδότηση, έχω εξετάσει πολλά σχέδια μεταρρύθμιση τη γη, εγγραφή ιδιοκτησία και προγραμμάτων χαρτογράφηση όλο τον κόσμο και εδώ θέλω να σα πω τι παρατήρησα και να προσπαθήσω να απαντήσω τι ερωτήσει αυτέ. Πρώτον, πρώτη παρατήρηση, πάντα θα είναι πολιτικά αμφιλεγόμενα τα δικαιώματα ιδιοκτησία, γιατί οι άνθρωποι πάντα ανταγωνίζονται λόγω τη έλλειψη πόρων. Αυτό θα είναι συνεχιζόμενο πρόβλημα. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και στα πλαίσια ε, διαμεσολάβηση για την επίλυση των συγκρούσεων. Πάντα θα υπάρχουν ε, προκλήσει στα υφιστάμενα καθεστώτα ε, δικαιωμάτων ιδιοκτησία, είτε πρόκειται ε, για, τους, ε, ε, για τα βοσκοτόπια έναντι της αγροτικής εκμετάλλευσης, είτε, για, είτε πρόκειται για ανάπτυξη αστικο, σε αστικές περιοχές, πρώην περιοχών της υπαίθρου κτλ. Τα περισσότερα προγράμματα δικαιωμάτων διοκτησίας δεν αντιμετωπίζουν τα βασικά ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι μικροϊδιοκτήτες στον αναπτυσσόμενο κόσμο και δεν υλοποιούν τα συστήματα τα οποία χρειάζονται οι πολύ φτωχοί για να, για να έχουν με, ε, με έναν τρόπο που είναι αποτελεσματικό σε πάψη κόστος πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα ιδιοκτησία. Αυτό προσπαθούμε να το επιλύσουμε χρησιμοποιώντα τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία ε, μειώνει δραστικά το κόστο εγγραφή, το κόστο συλλογή δεδομένων σε σχέση με τα αγροτεμάχια και στο ποιον ανήκουν κτλ. Ε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά όταν όταν έχουμε να κάνουμε ε, με τεμάχια τα οποία κοστίζουν η χαρτογράφησή του από 200 έως 1000 δολάρια το καθένα το κόστος χαρτογράφηση μπορεί να είναι το ίμιση τη αξία ε, συγκεκριμένη γη. Ε, αυτό δεν είναι εφικτό ε, ε, για οτιδήποτε και αν μιλάμε. Ε, να μην, ε, και να μην ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για πολύ φτωχέ περιοχέ. Άρα προσπαθούμε να μειώσουμε σημαντικά σε ένα λογικό επίπεδο, δηλαδή το κόστος εγγραφή. Και, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε GPS, χρησιμοποιούμε εικόνε δορυφόρου, χρησιμοποιούμε τεχνολογία η οποία έγινε διαθέσιμη σε εμά τα τελευταία 10 χρόνια. Και πραγματικά γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Γιατί έχουν αλλάξει βασικοί παράγοντε. Κάτι άλλο για το οποίο θα ήθελα να σας μιλήσω είναι για το πόσο ε, οι δωρητέ εστιάζουν την προσοχή του σε, σε παρεμβάσει από τα πάνω προ τα, προς τα κάτω. Αλλά αυτό ε, παραγνωρίζει ε, το γεγονό ότι τα δικαιώματα ιδιοκτησία συνδέονται άμεσα με την κοινότητα στην οποία αναφέρονται. Και επίση ε, τι ε, διεθνικέ, διεθνεί δηλαδή διαστάσει όσον αφορά τις, την ανασφάλεια του καθεστώτο ιδιοκτησία. Ποιο καθορίζει δηλαδή τα δικαιώματα ιδιοκτησία, όλα αυτά δημιουργούν ανασφάλεια και ασάφεια. Θα θεωρήσω λοιπόν εδώ ότι όλοι μας ζούμε σε ένα διαμέρισμα, σε ένα σπίτι. Και ότι όταν ε, μετακομίσατε συγκεκριμένο σπίτι, ε, έπρεπε να υπογράψετε ορισμένα χαρτιά τα οποία τα υπογράψατε και τα βάλετε σε ένα σιρτάρι. Όμως δεν είναι απλά χαρτιά αυτά τα οποία υπογράψατε. αποτελούν την εγγύηση της κυβέρνησης για το γεγονός ότι έχετε ορισμένα δικαιώματα στη συγκεκριμένη, ε, στο συγκεκριμένη οικία. Και είναι μια εγγύηση που στη Δύση είναι αξιόπιστη. Όμως αυτό είναι σχετικά το καινούριο. στις, στις ΗΠΑ ε, ε, ε, αυτό το δικαίωμα αποκτήθηκε μέχρι χρησικτησία Δηλαδή εγκαθίσαντο σε μια περιοχή και άρχισαν να την καλλιεργούν. Σιγά σιγά αυτά αναπτύχθηκαν σε οργανωμένες κοινότητες και τα δικαιώματα, τα δικαιώματα αναγνωρίζονται. Δηλαδή καταργούν τα παλιά δικαιώματα και αναγνωρίζονται τα δικαιώματα αυτών που κατέλαβαν τη συγκεκριμένη γη. Το γεγονό λοιπόν ότι έχουμε αυτά τα έγγραφα, τα οποία τα εγγυάται το, το κράτος, όλα αυτά είναι εμποδισμένα μέσα στο νομικό σύστημα. Αλλά αυτό είναι μειοψηφία γιατί οι περισσότεροι στον κόσμο δεν έχουν κανένα έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει την ιδιοκτησία του. Ε, και ορισμένοι ζουν με τη γνώση ότι μπορεί να του διώξουν από στιγμή σε στιγμή. Μία, ε, μία έκθεση των ΗΠΑ το 2003 ανέφερε ότι το 50% του πληθυσμού τη Καμπούλ στο Αφγανιστάν ε, ζούσε αντιμετωπίζοντα εντάλματα εκδίωξη από, από τα συγκεκριμένα σπίτια. Οι άνθρωποι λοιπόν είναι αναγκασμένοι να ζουν με αυτό that their property rights won't be respected. Ε, αντιμετωπίζουν λοιπόν ε, την απειλή τη έξωση διαρκώ. Σύμφωνα με του ερωτικού τομέα των δικαιωμάτων ιδιοκτησία, αυτή η ασάφεια ε, και η ανασφάλεια μειώνει το κίνητρο για επενδύσει, μειώνει την ικανότητα απόκτηση ε, χρηματοδότηση για να ξεκινήσει κάποιο την επιχείρησή του ή να, ε, σε, σε μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία ή να, ή να κάνει ε, συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει στο σπίτι του, αλλαγέ και τελικά ε, πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Πιστεύω λοιπόν ότι η θεωρία για τα δικαιώματα ιδιοκτησία είναι πάρα πολύ ε, σωστή. Γιατί αν δεν υπάρξει αυτή, ε, αν καταργήσουμε αυτή την ασάφεια, θα αλλάξουν οι ζωέ των ανθρώπων αυτών. Όταν δηλαδή θα έχουν βεβαιωμένα δικαιώματα ιδιοκτησία. Από τη δική μα την προνομιακή άποψη όμω εδώ στη Δύση, είναι εύκολο να ξεχάσουμε το πώ τελικά φτάσαμε σε αυτή την προνομιούχα θέση όπου η οικονομία της αγοράς είναι η κυρίαρχη μορφή της ανταλλαγής γης. Αυτή ε, ε, η εμπορευματοποίηση της γης και η ικανότητα ε, μέσω να, αγοράσει κανείς και να ανταλλάσσει τα, ακίνητα μέσω ε, ασφαλούς πίστης είναι σχετικά καινούρια. Ας πάμε λοιπόν λίγο πίσω για να δούμε πώς φτάσαμε στη μετάβαση, στη μετάβαση αυτή. Σε αναπτυσσόμενες χώρες λοιπόν όπου μεγάλο μέρος της γης είναι, δεν χρησιμοποιείται, όπου ε, το καθεστώς των ε, δικαιωμάτων είναι ανασφαλές. Ε, το γεγονός λοιπόν ότι καταλαμβάνουν ορισμένοι τη γη και αποκτούν δικαίωμα χρησικτησίας, αυτό είναι η βασική μέθοδος συνδιαλλαγής. Δεν πάει κανείς δηλαδή στην τράπεζα να πάρει ένα δάνειο για να αγοράσει ένα σπίτι. καταλαμβάνει ένα χωράφι, δεν ξέρει σε ποιον ανήκει, βλέπει ότι είναι άδεια, άδειο το χωράφι αυτό και το, το, το, το χτίζει τούβλο-τούβλο. Πώς δημιουργήθηκε λοιπόν το σύστημά μας και οι υποδομές για να φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Και πρέπει να δούμε και το πρόβλημα το οποίο ε, παρουσιάζεται εδώ. Το οποίο έχει να κάνει με το γεγονό ότι όταν εμεί κάνουμε εξαγωγή των αναπτυγμένων νομικών μα ε, συστημάτων στα πλαίσια τη αναπτυξιακή βοήθεια, τη ε, τεχνική βοήθεια προ αναπτυσσόμενε χώρε, εξάγουμε το τελικό προϊόν. Αλλά δεν εξάγουμε τα συστήματα, τα ενδιάμεσα. Όταν δηλαδή δημιουργούσαμε αυτή την αγορά. Όλα λοιπόν ε, τα σύγχρονα συστήματα αγοράς είναι το, ε, από το ιστορικό αποτέλεσμα αυτών των παραταμένων ε, διαφορών ανάμεσα σε, διάφορες, σε ομάδες διαφόρων συμφερόντων. Ε, όταν εμείς παρεμβαίνουμε στον αναπτυσσόμενο κόσμο, παίρνουμε το μέρος, ε, υποστηρίζουμε αν θέλετε το ένα από τα δύο μέρη της σύγκρουσης. Αλλά δεν έχουμε την ικανότητα να, να επιδείξουμε την απαραίτητη επιμονή, υπομονή Μερικές φορές ε, λοιπόν ε, ε, όλα αυτά είναι αποτελεσματικά, δηλαδή επιλύονται συγκρούσεις και δημιουργούνται αγορές. Αλλά μερικές φορές τα προγράμματά μας, παρόλο που τα φτιάξαμε με τις καλύτερες ε, προθέσεις, στην ουσία δημιουργούν ευκαιρίες για απάτες, για σφετερισμό και για, ε, και για, κατάληψη της γης. Βλέπουμε διαρκώς ότι τα εισαγόμενα νομικά συστήματα οδηγούν τελικά στην ομοποίηση της, της, της κλοπής και έτσι δημιουργούνται επαναστάσεις. Παράδειγμα, ε, η πολιτική, ε, η πολιτική στις, ε, στις Φιλιππίνες με την υποστήριξη των ΗΠΑ οδήγησε στην εξέγερση του Χουκ. η, χειρότερη περίπτωση κατά την άποψή μου είναι ότι καταλήγουμε στο να βοηθάμε τα κράτη τα οποία έχουν αποδείξει ότι είναι διεφθαρμένα και επεκτείνουν με αυτόν τον τρόπο την εξουσία, της, την εξουσία τους στις αυτο, αυτοδιοικούμενες κοινότητες όπως έκανε οι ΗΠΑ στο Βιετνάμ. Και σίγουρα αυτός είναι ο κίνδυνος σήμερα στο Αφγανιστάν. Πώς να δούμε λοιπόν, πώς θα δούμε το πρόβλημα αυτό και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των ιδιοκτήτων, ιδιοκτήτων γης που δεν έχουν το βασικό να καταλάβουμε εδώ είναι ότι υπάρχουν δύο είδη συγκρούσεων. Αυτά που αφορούν ε, του γείτονε, αν θέλετε, ε, τι ε, συγκρούσει οτίμων. Εκεί όμω το πρόβλημα επιλύεται είτε από του ίδιου του γείτονε, είτε από τι τοπικέ αρχέ. Το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων είναι ότι τελικά καταλήγουμε σε περισσότερη τεκμηρίωση και σε περισσότερη διαφάνεια αυτό που είναι διαφορετικό, ε, αυτό δημιουργείται για παράδειγμα ανάμεσα στις οικογένειες και, και είναι πιο κοινό στις οικογένειες. Εδώ έχουμε να κάνουμε τα ήθη, τα έθιμα ε, και όλα αυτά τα οποία είναι προβληματικά ακόμα και στον αναπτυγμένο κόσμο. Δηλαδή, μερικές φορές είναι, είναι, είναι συνηθισμένο να δημιουργηθούν ε, συγκρούσεις ανάμεσα ε, και στην ίδια οικογένεια. Και αυτό γίνεται ε, σε περίπτωση κληρονομιάς, ακόμα και σε βυτικό κόσμο. Ε, σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ε, και, και τι γίνεται. Όταν δεν ε, λειτουργεί η αγορά και δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και οι κληρονόμοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με τη γη αυτή, δεν μπορούν να την πουλήσουν. Ε, αυτό είναι ακόμα χειρότερο στην Αφρική, όπου για παράδειγμα πεθαίνει κάποιο και η οικογένεια του, δηλαδή τη γυναίκα του και τα παιδιά του, αντιμετωπίζουν έξωση από την υπόλοιπη οικογένεια. Αυτέ είναι τραγικέ συγκρούσει ε, μέσα στην ίδια την οικογένεια και, και, ε, και πραγματικά λύνονται με την παραδοσιακή προσέγγιση τη τεχνική βοήθεια, εκπαίδευση και τη νομική μεταρρύθμιση. Τα πράγματα διαφορετικά όταν πρόκειται για την εξουσία από το κράτο. Έχουμε ένα εξαιρετικό έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τίτλο Κατευθύνε γραμμέ για την πολιτική στον τομέα τη γη. Και αναφέρει ότι οι πολιτικέ αυτέ εκφράζουν τι πολιτικέ επιλογέ που γίνονται όσον αφορά την κατανομή τη ε, εξουσία ανάμεσα στο κράτο, στου πολίτε και τα τοπικά συστήματα ε, εξουσία. Πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε τα προγράμματά μα να μην αλλάξουν την κατανομή τη εξουσία και το σχετισμό των δυνάμεων υπέρ του κράτου. Ακόμα και όταν η έλλειψη ισορροπία δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αποτέλεσμα τη δική μα τη παρέμβαση, δεν υπάρχει μηχανισμό έτσι ώστε να αναλάβουν την ευθύνη για τη διαφθορά οι εθνικέ κυβερνήσει, για τι αυθαίρετε εξώσει ή για την πώληση των, φυσικών, των δικαιωμάτων φυσικών πόρων. Η διεθνή κοινότητα των δωρητών έχει την, ε, ε, πρέπει να δράσει με υπευθυνότητα. Ε, ιδιαίτερα λαμβάνοντα υπόψη ότι ε, σε πολλέ περιπτώσει, όταν πρόκειται για ασαφεί περιπτώσει, οι ιδιοκτήτε είναι πολυεθνικέ εταιρείε που έχουν την έδρα του στην Ευρώπη στι ΗΠΑ. Εμεί λοιπόν προσπαθούμε να σχεδιάσουμε φτιάσουμε ένα, ένα σύστημα με βάση τι χάρτε του Google για να αντιμετωπίσουμε το θέμα ε, των, προβλημάτων και τη εκδίκαση των διαφορών. Αλλά η καλύτερη λύση είναι να, προβλέψουμε τις, ε, τα προβλήματα πριν δημιουργούν. Εάν λοιπόν και οι μεγάλε πολυεθνικέ ήταν αναγκασμένε να εγγράψουν την, ε, γη που έχουν και τους φυσικούς πόρους και τι εκμεταλλεύσει φυσικών πόρων, τα πράγματα είναι διαφορετικά. με το κτηματολόγιο αυτό, με το μητρό αυτό, θα ενθαρρύνουμε την δημιουργία προτύπων σε διεθνέ επίπεδο. Και καθώ ε, συγκεντρώνουμε την εμπειρία μας αυτή και βλέπουμε την εμπειρία μας από όλες τις, από ε, τις ε, περιοχές βλέπουμε ότι απαιτούνται συγκεκριμένα δεδομένα για να έχουμε αξιόπιστα συστήματα παρακολούθησης. Και τα τελευταία 7 χρόνια αναπτύσσουμε αυτά, αυτό το σύστημα των βασικών προτύπων. Ε, και μέσα ε, στις προσεχείς εβδομάδες θα έχουμε και ένα ε, σχέδιο διεθνών προτύπων έτσι ώστε να έχουμε ένα διεθνές σύστημα για την τυποποίηση. Απαιτούνται πολύ περισσότερα για να εξασφαλίσουμε ότι είναι διαλειτουργικά τα διάφορα κτηματολόγια και να μπορούν να μεταφερθούν από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη τα διάφορα άτομα χωρίς να φοβούνται ότι θα υπάρξει σύγχυση για, το, για τα συγκεκριμένα τους δικαιώματα. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό ε, αυτού του, του Global Land Registry ε, θα ήταν, ε, είναι το γεγονός ότι μπορούν να υποβάλλουν τις απαιτήσει τους οι τοπικές κοινότητες και να ε, ε, κρατήσουν τα δικαιώματά τους, αν θέλετε, απέναντι σε περιπτώσεις κινδύνου. Θέλουμε να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα είδο εργαλείου ε, για να βοηθήσουμε με τη χαρτογράφηση και με την συλλογή στοιχείων, έτσι ώστε οι κοινότητες να αναλάβουν την ευθύνη για τα δικά του κτηματολόγια με τη βοήθεια βεβαίω μη κυβερνητικών οργανώσεων κτλ. Εργαζόμαστε με μία ε, με μια μη κυβερνητική οργάνωση ε, ε, στην Ινδία για να χαρτογραφήσουμε διάφορες περιοχές. Um, Και ε, ε, βεβαίω δεν θέλω να επιστρέψω στι τεχνικέ λεπτομέρειε, σα λέω όμω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το εγχείρημα αυτό. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να σα πω ότι ε, σήμερα το θέμα αυτό και η ιδιοκτησία θεωρείται ως ένα ε, βασικό και κυρίαρχο προνόμιο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, ε, αλλά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας είναι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία εξασφαλίζουν την επιβίωση του ανθρώπου, την ευημερία του και την ταυτότητά του. Ε, ο στόχο είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο ε, παγκόσμιο ε, οργανισμό που να μπορεί να πιστοποιεί και να προστατεύει τα δικαιώματα των μικροϊδιοκτητών. Βεβαίω δεν πρόκειται να τα λύσουν, το λύσουμε το πρόβλημα για πάντα, αλλά τουλάχιστον θα δώσουμε κάποια ανακούφιση σε αυτού των οποίων τα δικαιώματά του αμφισβητούνται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κλέιτον. Πολύ ενδιαφέρουσα η εισαγωγή αυτή που κάνουμε στη συζήτησή μα. Για να δούμε τα πράγματα στο σωστό του πλαίσιο, θα πρέπει να σας πω ότι δεν προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα πράγματα απλώς θεωρητικά και με αγαθές προθέσεις. Θέλουμε αυτή τη στιγμή να καταφέρουμε να συμβάλλουμε περισσότερο, να δούμε πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση τα τελευταία 20-30 χρόνια και πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις κακές πρακτικές. Οι άνθρωποι με τους οποίους εργάζεται ο Κλέιτον έχουν εκτιμήσει πάνω κάτω την αξία της μη κατεγραμμένης ιδιοκτησίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ακόμα και της παραγκουπόλεις, ακόμα δηλαδή και όλες αυτές τις κατοικίες για τις οποίες δεν υπάρχει κλιματολογιο ε, και η αξία κυμαίνεται από μερικά χιλιάδες δολάρια αναγροτεμάχιο μέχρι δεκάδες χιλιάδες δολάρια αναγροτεμάχιο και κατέληξαν στο συνολικό ποσό, στη συνολική αξία της μη καταγεγραμμένης ιδιοκτησίας παγκοσμίως. Το ποσό λοιπόν αυτό είναι 13 εκατομμύρια δολάρια. Ποσό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ε, έχουμε στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, της Φραγκφούρτης, του Λονδίνου συνολικά. Αν καταφέρουμε να περάσουμε την μη καταγεγραμμένη αυτή ιδιοκτησία, τη μη καταγεγραμμένη αυτή περιουσία σε κλιματολο σε ένα καθεστώς καταγεγραμμένης ιδιοκτησίας, θα καταφέρουμε να έχουμε τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να βγούνε από την οικονομική τους κρίση. Ακόμα και η Ευρώπη θα μπορούσε να βγει από την οικονομική της κρίση. Το πρόβλημα είναι ότι η ιδιοκτησία αυτή, η οποία δεν είναι καταγεγραμμένη, δεν μπορεί να τιτλοποιηθεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρηματοοικονομικά. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει ο Κλέιτον να βοηθήσει τους φτωχούς αυτούς ανθρώπους στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η οργάνωσή του. Θα ήθελα να καλέσω τώρα την Κλαρίσα Αγκουστίνους, που είναι επικεφαλής του τμήματος γης και διοκτησίας του UN Habitat, να πάρει τώρα το λόγο και να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, πώς μπορούμε να καταρτήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς για να έχουμε καλές πολιτικές για τη γη και την διοκτησία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέι Μίτσελ και τον κύριο Ντέβα για τη δυνατότητα που μου δίνουν να μιλήσω για τα δικαιώματα διοκτησίας, το καθεστώς διοκτησίας και την αρπαγή γης στις αμπτυσσόμενες χώρες. Επιστρέφω από μία συνάντηση με προσώπους της κυβέρνησης ε, του Ιράκ όπου ε, συζητήσαμε για το πώς θα καταφέρουμε να έχουμε στη χώρα αυτή μία πιο ανοιχτή αγορά, αποκεντρωμένη αγορά για την ιδιοκτησία, για την γη. Μία από τι βασικές προκλήσεις του 21ου αιώνα είναι να καταφέρουμε να απομακρυνθούμε από τις χαοτικέ πόλεις, οι οποίες θεωρούνται φυσιολογικές σε πάρα πολλέ χώρες του κόσμου και να πάμε τελικά σε μία βιώσιμη αστικοποίηση. Προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε μια καλύτερη διαχείριση της γη και της στέγασης. Εντολή του UN Habitat είναι η πρόθεση μιας κατάλληλης κατοικίας για όλους και μιας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και μπορούμε να δραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως καθότι το ίμιση της ανθρωπότητας ζει πλέον σε πόλεις και μέχρι το 2050 το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα κατοικεί σε αστικές περιοχές. Στις αναπτυσσόμενες χώρες η ανάπτυξη των πόλεων είναι πολύ μεγαλύτερη από τις συναπτυγμένες χώρες. Μάλιστα το 95% της αστικής ανάπτυξης παρατηρείται στις αναπτυσσόμενες χώρες και δυστυχώς βέβαια γίνεται με τη μορφή υποβαθμισμένων περιοχών μέσω φτωχογειτονιών και φτωσνικιών. Έχουμε 827 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στις συναπτυσσόμενες χώρες τέτοιες συνθήκες. Αν δούμε όμως τα πράγματα από την οπτική γωνία της ε, γης, θα δούμε ότι ε, ο χώρος που καταλαμβάνουν οι αστικές περιοχές αυξάνεται πολύ γρηγορότερα από ότι ο ίδιος αστικός πληθυσμός. Μεταξύ του 2000 και 2030 ο παγκόσμιος αστικός πληθυσμός θα αυξηθεί κατά 72%, ενώ οι οικοδομημένες περιοχές της πόλης θα αυξηθούν κατά 175%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μια τεράστια πρόκληση μπροστά μας όπως λέει και ο Πρόεδρος, για να καταρτήσουμε τα απαραίτητα αυτά εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να δώσουμε την απαραίτητη γη και στους φτωχούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει την σημασία της, των προτεραιοτήτων όσον αφορά την αστική ανάπτυξη και το 2009 είχαμε τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας για την κατοικία με βασικό θέμα τον σχεδιασμό του, αστικού μας μέλλοντος. Έλαβε χώρα λοιπόν μια τέτοια συνδιάσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συμμετοχή, μάλλον υπό την αιγίδα του Ευρωβουλευτή Μιγγελ Άγχελ Μαρτινές υπό την Προεδρία της κυρίας Εύα Ζολή και ε, με την παρουσία του κυρίου Γιάνν Όλμπριχτ, ο οποίος είναι επικεφαλής του ε, αστικού Intergroup του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέσω του UN Habitat έχουμε δώσει τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να βοηθήσουμε τις χώρες ΑΚΕ για την ε, εξυγίαση των υποβαθμισμένων περιοχών. Αν μιλήσουμε τώρα για την υγεία αυτή καθ' αυτή, όπως είπε και ο πρόεδρος, η κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντική η υγεία για να μας οδηγήσει στην απαραίτητη αυτή βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Και ουσιαστικά πειράζει πάρα πολλές πτυχές του πλανήτη μας σήμερα. Ο κλάδος όμως ανάπτυξης ε, της γης δεν έχει όλες τις απαραίτητες ε, όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να αντιμετωπίσει τι νέε προκλήσει. Και όπω μα είπε και ο προλαλή σα, γίνονται αυτή τη στιγμή κάποιε νέε διαρευνήσει. Πρέπει λοιπόν να καλύψουμε το κενό αυτό και να βρούμε τι απαραίτητε λύσει. Το UN Habitat προσπαθεί να διευκολύνει την ανάπτυξη του δικτύου GN Ενό δικτύου προκειμένου να καταφέρουν να απτυχθούν τα απαραίτητα εργαλεία. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό εταίρων οι οποίοι συνεργάζονται προκειμένου να καταλήξουν στα εργαλεία αυτά. Το δίκτυο αυτό το χρηματοδοτεί η Σουηδία και η Νορβηγία μέχρι στιγμή. Συμμετέχουν και άλλοι οργανισμοί όπω η IFAD, το Διεθνέ Ταμείο Γεωργική Ανάπτυξη, η ITC και η IHS που είναι ε, Ολλανδικά Ινστιτούτα Έρευνα και Κατάρτιση η ε, Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας, το Βασιλικό Ινστιτούτο των Τοπογράφων, το, η Ομοσπονδία των Γαλλόφωνων Τοπογράφων, η ΓΡΕΤ που είναι μια γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση, το ε, Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, καθώ επίση και το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί συνεργάζονται για την κατάρτιση αυτών των εργαλείων. Θέλουν λοιπόν όλοι αυτοί οι εταίροι να δημιουργήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να εφαρμοστούν πολιτικέ γη για του φτωχού και να γίνει απαραίτητη αγροτική μεταρρύθμιση όπου αυτό απαιτείται. Θέλουμε μια συνέχεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για όλους. Θέλουμε να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε μια διαχείριση της γης η οποία είναι ευνοϊκή για τους φτωχούς. Θέλουμε επίσης να καταφέρουμε να δώσουμε νέα όθηση σε κάποιες νέες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, το δίκτυο GLTN με την βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει βοηθήσει την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να δανειστεί 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να καταρτήσει ένα εθνικό κτηματολόγιο και ένα μητρό ακινήτων. Ένας άλλος στόχος είναι να βελτιώσουμε την, τον παγκόσμιο συντονισμό όσον αφορά τη διαχείριση της γης. Αναφέρομαι εδώ πέρα στην δήλωση των Παρισίων. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε πρόσφατη εμπειρία στην Κένια, όπου προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μία εναρμόνιση, μία ευθυγράμμιση και ένα συντονισμό της αναπτυξιακής βοήθειας όσον αφορά τον τομέα της γης και της ε, ιδιοκτησίας. Επίσης, στόχος επίσης του δικτύου είναι να βελτιωθεί η διάχυση και ανταλλαγή της γνώσης όσον αφορά την ασφάλεια της κατοχής γης. Χρησιμοποιώ τον όρο γη και όχι ιδιοκτησία, γιατί η ιδιοκτησία ουσιαστικά έχει να κάνει με την καταγεγραμμένη γη, την καταγεγραμμένη ιδιοκτησία. Και όπως σας είπα ήδη, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα περισσότερα αγροτεμάχια, το μεγαλύτερο τμήμα της γης στις αναπτυσσόμενες χώρες, περίπου το 70% δεν έχει περάσει κλιματολόγιο, δεν είναι καταχωρημένο σε μητρό. και περίπου ένα 2% μόνο ανήκει σε γυναίκες. Βλέπουμε ότι σε πολλά παγκόσμια προγράμματα για την γη δίνεται μία έμφαση όσον αφορά την χρησιμοποίηση των τίτλων ιδιοκτησίας και την προώθηση των τίτλων αυτών. Εργαζόμαστε όμως και αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή σε χώρες οι οποίες έχουν ένα μεγάλο επίπεδο ανισότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διαχειριστούμε και άλλα επιμερούς, ε, επιμερή ζητήματα, με συγχωρείτε, όπως ε, οι διάφορες διαμάχες που μπορούν να υπάρχουν γύρω από τη γη. Και αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά είναι ότι του τίτλου ιδιοκτησία χρησιμοποιεί συνήθω η πολιτική ελή ή οι πιο πλούσιε κοινωνικέ τάξει σε μια χώρα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτό το 70% το οποίο, το οποίο δεν είναι καταγεγραμμένο, βρίσκεται εκτός κλιματολογίου, επηρεάζει πάρα πολύ την ε, δημιουργία των ε, παραγκουπόλεων, την διαχείριση των πόλεων, την τοπική διακυβέρνηση και ουσιαστικά κατά επέκταση επηρεάζει και τις κλιματικές αλλαγές, την διατροφική ασφάλεια, καθώς επίσης και πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία μαστίζουν τον πλανήτη μας, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Και είναι πολύ πιθανό ότι η βιωσιμότητα του πλανήτη θα επηρεαστεί αν δεν αναπτύξουμε τα απαραίτητα εργαλεία και τις λύσεις που απαιτούνται προκειμένου να εφαρμόσουμε καλές πολιτικές για τη γη και την βιοκτησία. Οι εταίροι λοιπόν του GLTA εργάζονται για την ανάπτυξη των εργαλείων αυτών, αλλά έχουν πάρα πολλέ προτεραιότητε και χρειαζόμαστε πάρα πολλού εταίρου. Για παράδειγμα, ένα λονδικό πανεπιστήμιο ηγείται ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για την χρήση της γης και για την ανάπτυξη των απαραίτητων προτύπων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίω και για τους φτωχού πληθυσμού. Επίσης θέλουμε να εργαστούμε στην IT και για κάποια προβλήματα διαχείρισης τη γη, τα οποία μπορούν να προκύπτουν μετά από φυσικές καταστροφές. Επίσης πρόσφατα το GLTN με την βοήθεια του Πολωνικού Υπουργείου ε, διαχείριση τη γη Χωροταξία, διοργάνωσε μία συνδιάσκεψη για το ζήτημα αυτό. Καμία οργάνωση βέβαια και καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να δώσει τι απαραίτητε λύσει και μια μοναδική απάντηση σε όλα τα προβλήματα. Πρέπει να δούμε ποιε είναι οι κατάλληλε λύσει στα προβλήματα. Αυτό το οποίο υποστηρίζουμε είναι η πολιτική, η πρωτοβουλία διαχείρισης της γης που προωθεί, προωθούν τα Ηνωμένα Έθνη με την υποστήριξη της Αφρικανικής Ένωσης. Τον Ιούλιο του 2009 υποβλήθηκε η πρωτοβουλία αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να χρηματοδοτεί την εφαρμογή της πρωτοβουλίας αυτής. Συμμετέχει και το UN Habitat, ιδίως όσον αφορά την δημιουργία των απαραίτητων ικανοτήτων, το capacity building. Θα ήθελα τώρα να σας πω πώς μπορούν τα εργαλεία αυτά να ενδυναμώσουν τους επιτόπου πληθυσμούς. Πρόσφατα προσπαθούμε να καταρτήσουμε τα gender evaluation κριτήρια, τα κριτήρια εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν με την ε, αξιολόγηση της απόκτησης και χρήσης γης από το ένα φύλλο στο άλλο. Και θέλουμε να διαμορφώσουμε και τα εργαλεία προκειμένου να μπορούν να αποκριθούν στα κριτήρια αυτά. Και είδαμε ότι ε, καταφέραμε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αυτά να πείσουμε κάποιες τοπικές κυβερνήσεις που προσπαθούσαν να κάνουν έξωση σε κάποιους τοπικούς πληθυσμούς να αλλάξουν την άποψή τους, να μην εκτοπίσουν τους πληθυσμούς αυτούς και μάλιστα να αναβαθμίσουν τις ε, γειτονιές στις οποίες ε, ζουν. Προκειμένου να συνδέσω το ζήτημα αυτό με το επόμενο πάνελ, θα ήθελα να σας πω ότι ε, χωρίς τα νέα αυτά εργαλεία διαχείρισης της γης δεν είναι δυνατό για πάρα πολλές χώρες να καταφέρουν να εφαρμόσουν βιώσιμες πολιτικές αστικοποίησης και δεν θα καταφέρουν να φτάσουν ούτε στην καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση ούτε στην εξάλληψη της φτώχειας. Είναι πολύ σημαντικά τα εργαλεία αυτά για την καλύτερη δυνατή διακυβέρνηση και για να καταφέρουν να ρυθμίσουν καλύτερα την ανεξέλεγκτη απόκτηση γης όπως αυτή συμβαίνει σήμερα σε πάρα πολλές συναπτυσσόμενες χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα σειρά παρατηρήσεων. Τώρα, ο επόμενος ομιλητής ε, που θα μας δώσει κάποια πρακτικά παραδείγματα το τι ε, ε, θα μπορούσαν να κάνουν και έκαναν και η ομιλήτρια και η εταιρεία της στη Ρουάντα. Ξέρετε τι φρικτή εποχή πέρασε η Ρουάντα. Τώρα η κατάσταση είναι σταθεροποιημένη, βρίσκεται στο δρόμο τη ανάπτυξη; άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ε, εταίρους, ε, γιατί stakeholders, γιατί ε, είναι πολύ σημαντική για την προστασία της γης. Αν δεν έχουν τίποτα να προστατεύσουν, ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Καλό λοιπόν την Unlock να πει δύο λόγια για την εργασία στη Ρουάντα. Thank you. Um... Σας ευχαριστώ. Βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για την ε, επίσημη διαδικασία ε, τίτλοποίησης ε, στην δημιουργία τίτλων στην Ρουάντα. Αρχικά με χρηματοδότηση από το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση και στη συνέχεια από άλλα μέσα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για την οποία η εταιρεία μου, η TSP, έχει αναλάβει τη διαχείριση. Βρισκόμαστε ε, στην πιλωτική φάση τώρα, σε και, ε, τελειώσαμε την πιλωτική φάση και είμαστε δεύτερη φάση σε πανεθνικό επίπεδο. Γιατί στη Ρουάντα. Λοιπόν, ε, η Ρουάντα πραγματικά είναι εμβληματικό πρόγραμμα και όσον αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, ε, που είναι συμμετοχική και χαμηλού κόστους, και λόγω του επίπεδου δέσμευσης και της κυβέρνησης αλλά και του λαού, των πολιτών της Ρουάντα απέναντι στο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι μερικέ φορέ να κατανοούμε γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, για παράδειγμα τη Ρουάντα, αποφάσισε να ακολουθήσει την οδό ε, της επίσημης δημιουργίας τίτλων. Όταν τα τελευταία 7-8 χρόνια ε, από τότε δηλαδή που η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε το έγγραφό της για την ιδιοκτησία της γης, 2003, ε, και στη συνέχεια ε, υπήρξαν οι κατευθυντήριε γραμμέ για την πολιτική γη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε ε, αυτό ο προβληματισμό και αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη σημασία για την αναγνώριση δηλαδή των συστημάτων ε, εθνική κατοχή γη. Να σα πω λοιπόν γιατί η κυβέρνηση τη Ρουάντα αποφάσισε να ακολουθήσει την πιο επίσημη διαδικασία απονομή τίτλων. Θα μιλήσω για την νομική βάση, για τη θεσμική βάση όσον αφορά αυτό το νέο σύστημα και το πρόγραμμα, γιατί δεν πρόκειται για κάτι το οποίο έγινε έτσι τυχαία και σπασμωδικά. Και στη συνέχεια θέλω ήθελα να πω δύο λόγια, στον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, το πώς αυτή η διαδικασία τίτλων ε, αναπτύχθηκε και να σας μιλήσω για τη μεθοδολογία. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Εν μέρη διότι όλα αυτά ε, έχουν να κάνουν με την ίδια την επιτυχία του προγράμματος και επειδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα προσδιορίζουν, ε, θα προσδιορίσουν το πόσο σημαντική θα είναι η εμπειρία της Ρουάντα και της άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Θα, προσπαθήσω να βγάλω αυτό το μικρό κουτάκι που λέει PDF complete από την οθόνη σας. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω. Σας ζητώ συγγνώμη. It's at the top. Sorry about that. I, can read it. It's just a... Δεν είναι ότι εγώ δεν μπορώ να διαβάσω. Μάλλον ε, είναι ενοχλητικό για εσά. Τέλο πάντων. Λοιπόν, αν ε, μπορώ, μου επιτρέπετε να αρχίσω ε, από την αρχή, να σα πω πώ ξεκίνησε το πρόγραμμα και μέσα στα πλαίσια, και τα πλαίσια μέσα στα οποία αναπτύχθηκε. Η Ρουάντα μετά από την γενοκτονία του 1994 Μέχρι το 1999 βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Ε, είχαμε την επιστροφή των πρόσφυγων, ε, τα εσωτερικά εκτοπιστέντα άτομα τα οποία γύρναγαν στον, τρόπο, στον τόπο καταγωγή του. και η κυβέρνηση επέλεξε του τους μηχανισμού σε κάθε ε, περιοχή. Προσπάθησε λοιπόν να βοηθήσει με τον τρόπο αυτό την επίλυση των διαφωνιών όσον αφορά την κατοχή τη γη. Μετά το 1999 προσπάθησαν να ακολουθήσουν μια πιο δομημένη ε, και πιο επίσημη προσέγγιση για τα ζητήματα της γης και ξεκίνησε η συζήτηση για την πολιτική γης και για την νομοθεσία που απαιτείται για την επίλυση των, διαφόρων, ε, των επιμέρους διαφορών. Και τότε άρχισε να προκύπτει η ανάγκη για μια επίσημη πολιτική στον τομέα της ιδιοκτησίας. Η κυβέρνηση θεώρησε λοιπόν ότι ε, η κοινωνική δομή και το εθιμικό δίκαιο είχε καταρρεύσει. Δηλαδή πριν την γενοκτονία υπήρχε η έξοδος από το 1959, έξοδος των ανθρώπων. Ε, θεωρούσαν λοιπόν ότι οι φυστάμενε δομέ δεν υπήρχαν ότι οι προηγούμενε δομέ δεν υπήρχαν και δεν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ε, την επίλυση διαφορών ή αναγνώριση ε, δικαιωμάτων ιδιοκτησία, ενώ αυτό το είχαν πετύχει στο παρελθόν. Επίση η αναγνωριση θεώρησε ότι ε, το εφιστάμενο σύστημα, το προηγούμενο σύστημα, είχε ορισμένε ιδιότητε που συνέβαλαν και στον πόλεμο και στη σύγκρουση. Άρα λοιπόν ήρθε η στιγμή, θεώρησε η κυβέρνηση, να σταματήσει το σύστημα αυτό. Μπορεί επίση να υπήρξε και κάποια επίδραση ε, των ε, δωρητών από τη Δύση. Γιατί η χώρα αυτή τότε ήταν εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από τις δωρεές. Πρόκειται λοιπόν για μια νομική και θεσμική βάση. Και ε, αυτό πραγματικά κατέστησε αυτή την πολιτική πιο συστηματική. Το 2004 ανεκρίθη η πολιτική γης που είχε αναπτυχθεί με συμμετοχικό τρόπο με τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Και οι δύο βασικές αρχές αυτής της πολιτικής ήταν η ισότητα και η ασφάλεια, η εξασφάλιση της πρόσβασης στη γη και η διαρκής και βέλτιστη ε, χρησιμοποίηση της γης και, της, και ανάπτυξη και η καλά καθορισμένα, ε, ε, ε, ένα σωστά καθορισμένο και ενισχυμένο θεσμικό και νομικό πλαίσιο θεωρήθηκε ως ουσιαστικό για την υλοποίηση πολιτικής πολιτικής. Και στη συνέχεια είχαμε την έγκριση της επίσημης νομοθεσίας του Οργανικού Νόμου για τη Γη το Νοέμβριο του 2005, που περιείχε τρία βασικά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο ήταν ότι καταργήθηκε το εθνικό δίκαιο ιδιοκτησίας, παρόλο που προστατεύονταν οι πρώην ιδιοκτησίε. Δεύτερον, ε, ένα σύστημα υποχρεωτικό σε πανεθνικά πλαίσια. Επίση, επιβεβαιώθηκε ε, η φύση των δικαιωμάτων ε, γη και εκτό από ένα μικρό ποσοστό γη το οποίο ήταν χαρακτηρισμένο από ιδιωτικά δικαιώματα ε, γης ε, που είχαν κληροτηθεί από το παλιό επικοινωνικό σύστημα. Ε, τα υπόλοιπα ήταν κρατικής ιδιοκτησίας που είχαν εκμισθωθεί μέσα από μακροχρόνια μισθωτήρια συμβόλαια από το κράτος για 15 έως 19 χρόνια. Ε, δηλαδή, από τη μια όμως είχαμε την, ε, ε, τη δημόσια κατοχή αυτών των, αυτή, αυτής της γης και από την άλλη υπήρχε μια ολόκληρη ιδιωτική αγορά, αν θέλετε, αγοραπολισίας αυτών των μισοτηρίων συμβολέων. Τώρα, να σας πω λίγο περισσότερα... Να σα δώσω λίγο περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα καταχώρηση, το πρόγραμμα εγγραφή κτηματολογίου. Το πρώτο που έγινε ήταν ε, να, δημιουργηθούν, να δημιουργηθεί μια σειρά νέων θεσμών και δομών ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να είναι ξεκάθαρε οι υποχρεώσει και οι αρμοδιότητε του κάθε θεσμού. Όπω ακούσαμε και από τι προηγούμενε ομιλίε, μερικέ φορέ η νομοθεσία είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν εφαρμόζεται σωστά, διότι έχουμε επικαλυπτόμενου ρόλου και αρμοδιότητε ή συγκρόμενου ρόλου. Και βεβαίω δεν έχει επιληθεί απόλυτα το πρόβλημα αυτό στη Ρουάντα, αλλά σίγουρα αντιλήφθηκε η κυβέρνηση ότι ε, έπρεπε να υπάρχουν θεσμοί που να είναι απευθεία αρμόδιοι για την εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία. Από το 2006 μέχρι το 2009 υπήρξε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα σε τέσσερι ε, περιοχέ. Ε, δεν κάλυψε και, τις πέντε, και τους πέντε νομούς αν θέλετε, αλλά τις τέσσερις. Και εκεί προσπαθήσαμε να δούμε κατά πόσον αυτή η αποφασιστική κίνηση της κυβέρνησης θα ε, ξανάνοιγε παλιέ πληγέ κτλ. Γιατί κοιτάξτε, αυτό ήταν ο βασικό φόβο τη κυβέρνηση. Άρα είχα, υπήρχαν ήδη δύο στόχοι έναντι του πιλωτικού σχεδίου. Το πρώτο είναι να ελέγξουμε τη μεθοδολογία και να είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά θα οδηγούσε στου ευθέου στόχου. και απ' την άλλη να δούμε κατά πόσον ε, οι πολίτε ήταν έτοιμοι να δεχθούν το καινούριο σύστημα και να, είμαστε, να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργούσε, δημιουργούσε Πάντω γενικά πρέπει να σας πω ότι ήταν ευρύτερη αποδοχή από, τον, ε, από τους ανθρώπους, από το λαό της Ρουάντα. 15.000 αγροτεμάχια ε, καταχωρήθηκαν καλύπτοντας ε, μια συνολική ε, επιφάνεια 3.500 εκταρίων. Και αυτό που ε, είναι ενδιαφέρον είναι ότι ήταν πολύ ε, μικρό το ποσοστό των ε, προβλημάτων και των διαφωνιών. Και λαμβάνοντα υπόψη την ιστορία τη Ρουάντα, αυτό ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστο. Και οι διαφωνίε αφορούσαν κυρίω την ίδια την οικογένεια. Αυτό το είπε και ο Κλέιτον. Είναι αρκετά συνηθισμένο να υπάρχουν ενδοοικογενειακέ διαφορέ. Σε αυτή τη διαδικασία επίση δημιουργήθηκε και η θεσμική υποδομή και ενισχύθηκε. Η δεύτερη φάση ε, που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι ε, η αναβάθμιση αυτής της πιλωτικής ε, φάσης σε εθνικό επίπεδο. Και βεβαίως υπήρξαν ορισμένε δυσκολίε με τη χρηματοδότηση, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να ε, κρατήσει τις δομές που δημιουργήθηκαν στο πιλωτικό ε, σχέδιο με στόχο την οριοθέτηση 800.000 αγροτεμαχίων μέχρι το τέλος ε, του Ιουνίου 2010. Δηλαδή ένα πρόγραμμα με πολύ ψηλότερους στόχους, αλλά, αλλά κοιτάξτε, ένα ε, συνολικά μέχρι το 2012 είναι 8 εκατομμύρια ε, αγροτεμάχια. Καταλαβαίνετε λοιπόν είναι πάρα πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι βεβαίω κατά πόσον ο στόχο αυτό ε, θα επιτευχθεί απόλυτα και κατά πόσον η προβλέψει είναι ακριβεί. Τώρα, θα σα πω δύο λόγια για αυτή τη μεθοδολογία. Βλέπετε ένα διάγραμμα ροή που μάλλον είναι δύσκολο να το διαβάσετε. Θα σα το εξηγήσω. Θα σα πω δύο λόγια για τα πρώτα βήματα και μετά θα σα δείξω ορισμένε εικόνε που μιλούν από μόνε του. Για να καταλάβετε το πώς γίνεται αυτή η εγγραφή στο κτηματολόγιο. Πρώτα απ' όλα, εντοπίζονται οι περιοχέ στι οποίε θα γίνει η εγγραφή, ειδοποιούνται έγκαιρα οι κάτοικοι, γίνεται εκστρατεία ενημέρωση, ευαισθητοποίησης, ε, ε, ε, γίνεται η συζήτηση, εκφράζουν αντιρρήσει του, τα πιθανά ωφέλη και μετά έχουμε τις ε, τοπικές αρχές ε, που ε, κάνουν την, την εγγραφή. Δηλαδή γράφουν σε κάνουν εγγραφή σε ένα βιβλίο, δίνουν μια απόδειξη ε, ε, όπου ο κάτοχος ε, ε, ζητά δικαιώματα στην περιοχή αυτή. Λοιπόν, να δείτε τι γίνεται με την οριοθέτηση. Είναι μια ιδιαίτερα κοινωνική δραστηριότητα. Βλέπετε αυτούς τους, πόσοι πολλοί είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι περπατούν κατά μήκο τη οριοθέτηση. Αυτή τη μεθοδολογία χρησιμοποιούμε. Δεν χρησιμοποιούμε παραδοσιακές μεθόδους χρησιμοποιούμε ε, δορυφορικές ε, εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Όπως είπε και ο Κλέιτον, η τεχνολογία μας βοηθάει ιδιαίτερα γιατί έχει εξελιχθεί. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους ε, δορυφορικούς χάρτες ε, που αφορούν ολόκληρη την χώρα με κλίμακα ένα προς 2.000 στις αγροτικές περιοχές και ένα προς 1.000 στις ε, αστικές περιοχές. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ δεν χρησιμοποιούμε ε, ερευνητές ε, επαγγελματίες, αλλά ανθρώπους, κατοίκους που γνωρίζουν πολύ καλά τη συγκεκριμένη περιοχή και που μπορούν να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά που βλέπουν στο χάρτη και να εντοπίσουν τα, τα όρια με τους ιδιοκτήτες. Περπατούν δηλαδή τα, ε, κατά μήκο των ορίων με τους ιδιοκτήτες, με τους γείτονες. Όλοι δηλαδή ε, οι εμπλεκόμενοι συμμετέχουν και με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος απάτης ε, ή ε, ψευδών ισχυρισμών. Όπως βλέπετε εδώ, όλοι ε, βρίσκονται πάνω από το χάρτη και βλέπουν τη χάραξη των συνόρων και εκφράζουν την ικανοποίησή του σημεί. Μετά πηγαίνουν το αποτέλεσμα στην τοπική επιτροπή, καταγράφουν τη, συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία και δίνουν την απόδειξη για τον ισχυρισμό του τίτλου με... και μετά έχουμε κάποια ενδιάμεσα βήματα μέχρι να δοθεί ο επίσημος τίτλος. Υπάρχει βεβαίως και η επίσημη ανάθεση εκεί όπου επιλύονται και οι διαφορές αν υπάρχουν. Το πρώτο επίπεδο είναι ε, το αμπούντζι, δηλαδή ε, το τοπικό συμβούλιο του, του χωριού. Εάν δεν μπορεί να επιληθεί η διαφορά σε αυτό το επίπεδο, ε, πηγαίνει στο επόμενο, που είναι το παραδοσιακό δικαστικό σύστημα. Αλλά αυτά γίνονται σε πολύ μικρό βαθμό. Βέβαια, το τονίζω ότι βρισκόμαστε στην πιλωτική φάση. So what are some... Να δούμε λοιπόν ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν σε αυτή τη διαδικασία καταχώρησης. Ξεκινώ με το πρώτο υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην οριοθέτηση, δηλαδή στον ε, επιτόπου καθορισμό των συνόρων και στη χάραξή του στο χάρτη, μέχρι ε, την επίσημη έκδοση του τίτλου. Η οριοθέτηση προχωράει ιδιαίτερα γρήγορα, οι δομέ έχουν δημιουργηθεί και τελικά έχουμε συμφόρηση ε, στι υπηρεσίε έκδοση τίτλων. αυτό καταλαβαίνετε ότι ε, είναι ένα πρόβλημα, γιατί μπορεί σε τελευταία ανάλυση να υπονομεύσει ε, το σύστημα και, την, ε, και το γεγονό ότι οι άνθρωποι θα χάσουν την εμπιστοσύνη του στο σύστημα. Αν δεν πάρουν τον τίτλο του, τότε τελικά πρέπει να χάσουν την εμπιστοσύνη του. Ε, και τελικά να γίνονται αγοραπολισίε με βάση αυτά τα ανεπίσημα χαρτιά εγγραφή, ε, τελικά να υπάρξει πρόβλημα και να την αφήσει στον αέρα το σύστημα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν δύο σημεία ε, όπου, όπως σας είπα, παρουσιάζεται συμφόρηση. Το ένα, συμφόρηση. Το ένα είναι διοικητικό, δηλαδή απαιτούν προσφέρει ε, για να επεξεργαστούν αυτά, αυτές τις προσωρινές αποδείξεις, να ε, καταχωρήσουν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα όρια κτλ. Ένα άλλο σημείο συμφόρησης βρίσκεται εκτός του ελέγχου μας είναι, και αφορά το ίδιο το δικαστικό σύστημα. Αν αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των ε, διαφορών, ακόμα και αν σε απόλυτους όρους, ακόμα και αν ε, σε ποσοστιαίους δεν ε, αυξάνεται ο ρυθμός αυτός, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δούμε τις δυνατότητες του δικαστικού συστήματος. Δεν θέλουμε συμφόρηση στα δικαστήρια, θέλουμε να επιλύονται γρήγορα διαφορές αυτές. Ένα άλλο ζήτημα είναι ποιος αναλαμβάνει το κόστος της τιτλοποίησης έκδοσης τίτλων και σε ποιο επίπεδο. Η κυβέρνηση της Ρουάντα πιστεύει ότι ε, πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή οι πολίτε ε, πρέπει να πληρώνουν για την παροχή υπηρεσιών και δεν θέλει να επαναχωρήσει από αυτή την αρχή. Εδώ όμω υπάρχει ε, και ένα είδος μικτής χρηματοδότησης ανάμεσα στην Ήπεθρο και στις αστικές περιοχές. αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το κόστος είναι πολύ χαμηλό λόγω της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε γιατί ε, χρησιμοποιούμε την ε, ε, τεχνολογία, την άκρως εξελιγμένη τεχνολογία που τώρα είναι διαθέσιμη και φθηνότερη, χρησιμοποιούμε τους τοπικούς κατοίκους, άρα δεν έχουμε όλα αυτά τα διοικητικά κόστη. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Ε, συμμετέχουν ιδιαίτερα οι πολίτες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να εργαστούν είτε θελοντικά είτε με ένα συμβολικό αντίτιμο. Όλοι λοιπόν συνέβαλαν και συμβάλλουν σε αυτό το πρόγραμμα έκδοση τίτλων, το οποίο είναι πολύ χαμηλού κόστου. Εξακολουθεί όμω να υπάρχει ένα κόστο και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για πολύ φτωχού ανθρώπου. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτηση. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η, ε, η διαδικασία αυτή και τι διδάγματα μπορούν να αντιληφθούν για άλλε και τι υπόλοιπε χώρε. Το γεγονό ότι είναι χαμηλού κόστου είναι σημαντικό. Αλλά μπορεί να μην είναι τόσο ακριβές ε, όσο οι παραδοσιακές κλασικές ε, διαδικασίες οριοθέτησης. Και αυτά πρέπει να τα ζυγίσει κανείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις ε, όπου είναι πολύ, έχουμε πολύ σημαντικές διαφορές, τότε εκεί μπορεί να απαιτούνται πιο αξιόπιστα στοιχεία. Άρα ε, αυτά ε, στη φάση του σχεδιασμού θα πρέπει να σκεφτεί κανείς πολύ καλά ε, πριν αποφασίσει ότι θα μεταφέρει τη μεθοδολογία της Ρουάντα και στις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης θεσμική ρόλη και δυνατότητα για διαδικασίες καταχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας μεγάλης κλίμακας. Σας το είπα, βρισκόμαστε στο πιλωτικό σχέδιο και η πρόκληση είναι πολύ υψηλή ε, όταν μιλάμε για πανεθνική εφαρμογή του προγράμματος μέσα σε δύο χρόνια. Παρακολουθούμε λοιπόν στενά ε, το, ε, το ζήτημα των θεσμών και τι είδους προσαρμογές πρέπει να γίνουν. Εξακολουθεί να υπάρχει μια έλλειψη αντιστοιχία ανάμεσα στα επίσημα νομικά συστήματα, τα οποία είναι πιο προσαρμοσμένα με τη βυτική ε, κουλτούρα ε, και διαφορά λοιπόν και έλλειψη αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό ε, και στο, στα συστήματα θυμικού δικαίου, τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν. Παράδειγμα, στη Ρουάντα απαγορεύεται η πολυγαμία επίσημα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει στην πράξη. Πώ αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα σα πω και κάτι άλλο. Έχουν βρει, ε, είναι ιδιαίτερα εφευρετικοί οι άνθρωποι ε, και βρίσκουν τρόπους και ξεφεύγουν. Αλλά αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ορισμένες εντάσεις σε ορισμένε περιπτώσει και όσον αφορά την ιδιοκτησία. Και επίση κάτι άλλο. Πώ μπορεί κανεί να, να, δημιουργήσει τα κατάλληλα συστήματα και τι κατάλληλε δομέ για την διατήρηση ενό συστήματο κτηματολογία εν ώψη των συναλλαγών. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Ε, για οποιοδήποτε πρόγραμμα ε, πρώτη εφαρμογή κτηματολογίου, αν κανεί δεν μπορεί να το διατηρήσει βιώσιμο και να εντάσσει όλε τι συναλλαγέ, δεν έκανε τίποτα. Και αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μόλι σκέφτεστε ε, για την δημιουργία αυτού του προγράμματο, αυτό πρέπει να το έχετε στο μυαλό σα. Άρα, τελειώνω εδώ τελευταίες τρεις παρατηρήσεις που ήδη σας τα είπα. Η μεθοδολογία στη Ρουάντα αποτελεί ένα καλό σημείο αναφορά για ε, έκδοση τίτλων ιδιοκτησία χαμηλού κόστου στην, στην Αφρική και σε άλλε αναπτυσσόμενε χώρε, αλλά θα πρέπει ε, να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερε συνθήκε κάθε χώρα και πάντα να εξετάζεται η ισορροπία ανάμεσα στι κοινωνικέ και πολιτικέ προτεραιότητε και στο κόστο. Ε, Πάντω, ε, κοινωνικέ και πολιτικέ προτεραιότητε και η υποστήριξη των ανθρώπων είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σα ευχαριστώ. Very... Σα ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμε αυτέ τι πληροφορίε που μα έδωσε για τι επιτόπου εμπειρίε που είχατε. Όταν φτάσουμε στι ερωταποκρίσει, θα έχετε σίγουρα πάρα πολλέ ερωτήσει. Αναφερθήκατε σε 8 εκατομμύρια αγροτομάχια. Πόσο θα κοστίσει, πέστε μου αργότερα. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω την Ελέν Ροσκούτ, τον Αλέν Ροσκούτ να μου λύσει για τη δική του εμπειρία ως μέρος Τεχνικής Επιτροπής ε, για την ε, κτίση της γης στην Μαδαγασκάρη και να μας πει πώς οι δικές του εμπειρίες είναι παρόμοιες ή διαφορετικές από τις ε, εμπειρίες της Άννας. Eh bien, paradoxalement, elle n'est pas fondamentalement différente. Όχι, οι δικέ μου εμπειρίε δεν είναι ουσιαστικά διαφορετικέ και μάλιστα προηγουμένω που συζήτησα με την Άννα, ήθελα να σα πω ότι στα τέλη τη δεκαετία του 90 και αρχή τη ε, δεκαετία του 2000 γνώρισα την ε, κατάσταση στην Ρουάντα όταν τότε προετοιμάζονται μια καινούρια ε, πολιτική. Μία εικόνα θα υπάρχει στην δική μου παρουσίαση, το οποία θέλω να επιστήσω την προσοχή σας. Καταρχήν, το διαφοροποιημένο του, ε, του τοπίου. Ε, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ε, ε αγροδομαχίων, πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος της καταγραφής ε, των ε, αγροτομαχίων αυτών, καταλαβαίνετε, βλέπετε την εικόνα, το να χρησιμοποιήσει κανένας εδώ μια μέθοδο για να ε, μπορέσει να βρει τα όρια αυτών των ε, αγροτομαχίων, είναι πάρα πολύ ακριβό, να χρησιμοποιήσει οι κόρες από δορυφόρους πάλι είναι πολύ ακριβό. Έχουμε λοιπόν προβλήματα τεχνολογίας και κόστους. Υπάρχει και ένα νομικό πρόβλημα όμως επιπλέον. Αναφέρθηκε το νομικό πρόβλημα όταν αναφέρθηκε ο Φερνάντο Τεσότο, ο οποίος ήδη ανέφερε κάποια προβλήματα για το κεφάλαιο και είπε ότι τα πραγματικά προβλήματα των χώρων αυτών είναι ότι οι εργασίες γίνονται από ντόπιου νομικούς αλλά που χρησιμοποιούν ε, χρησιμοποιούν όμως εξωτερικούς νομικούς που δεν γνωρίζουν την τοπική κατάσταση Μεταρρύθμιση λοιπόν που υπάρχει εδώ και το 2007 είναι η λεγόμενη προπριετέ γκάσιο. Δηλαδή είναι η διοκτησία των σελίτ, των προχόντων, εκείνο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ε, αστικό κώδικα της Γαλλίας και το σύστημα Torrents επίσης Αυστραλιανό δηλαδή νόμο του 1850. Ε, και τώρα τελευταία έχει στη Μαδαγασκάρη ένα καινούριο σύστημα που βασίζεται στην ε, πολιτισμό της Μαδαγασκάρης και τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται το δίκαιο στη χώρα αυτή. Και πραγματικά δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά. Δεν μιλάω πολύ καλά τη γλώσσα, αλλά δεν υπάρχει μια λέξη που να λέει ιδιοκτησία, που να λέει εγώ είμαι ιδιοκτήτη γης. Υπάρχουν διάφορες λέξεις που χρησιμοποιούνται ανάλογα με το, τη χρήση που γίνεται της ε, γης, ανάμεσα με τις δυνατότητες μεταβίβασης στην οικογένεια και ο καθεξής. Τονίστηκα προηγουμένως, θα το περάσω σαν γλίγορα, γιατί παίζει και εδώ το ρόλο του, η σημασία της, ε, του ελέγχου αυτού της, ε, της Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ό,τι και να κάνει κανένα βρίσκεται μέσα στα πλαίσια τη έκθεση για τα αγροτεμάτια. Όπου και να βρίσκεται, είτε κατοικεί μέχρι και να φτάσει στο νεκροταφείο. Εγώ εργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια, από το 1970, έμαθα επιτόπου στην Αφρική, πράγματα που δεν ήξερα καθόλου. Εγώ ήξερα νόμιζα τα πάντα με τις υποθήκες, με το άρθρο 644 του κώδικα, αλλά εδώ έχουμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα, την οποία ανέφεραν όλοι οι προλαλήσαντες. Δηλαδή υπάρχει μία μη αποκλειστικότητα της ε, ε, ε, με την έννοια της επιφάνειας. Όμως στις πολιτισμούς αυτούς του Νότου υπάρχει μια πολύ πιο πλούσια εικόνα. Δηλαδή υπάρχουν για την ίδια επιφάνεια διαφόρου τύπου δικαιώματα ιδιοκτησίας. Αυτό που ελέγχθη. Όταν φτάνουμε οι ιερείς στις... Ε, ε, όταν φτάνουν οι βοσκοί στα, στα χωράφια όπου είχε καλλιεργηθεί το ρύζι, μετά που θα είχε κοπεί το ρύζι στη Μαδαμασκάρη, δεν έρχονται χαριστικά, αλλά γιατί έχουν και εκείνοι ένα πραγματικό δικαίωμα ιδιοκτησίας για τη γη αυτή. Αυτή η έννοια που εμείς ε, στις, ε, στους δικούς μας πολιτισμούς ε, δίνουμε στην ιδιοκτησία, όχι της χρήσης ή της χρησιμότητας τους γης, αλλά της ε, επιφάνειας της γης αυτής είναι διαφορετική. Το σύστημα Torrents έχουμε εκεί, δηλαδή κατά τη διάρκεια της γαλλικής ε, απεικιοκρατής περιοχής, ε, εποχής, θεωρείται ότι υπήρχε ε, κάτι πολύ πιο σύγχρονο. το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, όπως το έχουμε εμείς, είναι σαν μια Rolls που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως παντού. Οι τίτλοι, οι τίτλοι ιδιοκτησία της γης, δηλαδή τα κτηματολόγια, δεν προβλέπουν μόνο την καταγραφή, δεν θα είχε νόημα. Υπάρχει αφενός, αφενός καταγραφή, δηλαδή οριοθετώ ένα αγροτεμάχιο. Οι μέτρες το κάνουν αυτό πολλές φορές από το κράτος. Καμιά φορά είμαστε εγκεκριμένοι από το κράτος. Είναι εκεί πάντα δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Ο πρόεδρος είπε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Λοιπόν, εδώ και μερικά χρόνια ήμουν στο Ιμπεργοβούλ, μεταξύ Μαλέν στο νέο αεροδρόμιο και το... την πρωτεύουσα. Έπρεπε να τα γράψουμε όλα τα αγροτομάχια. Τα προβλήματα που γνωρίζουμε είχαν καταγραφεί από τους ε, εκπροσώπους του κτηματολογίου που όταν πήγαιναν να καταγράψουν ένα αγροτεμπάχιο ζητούσαν 30% για συμπληρωματικό κόστος ας πούμε. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να ανοιχθευτεί η επιφάνεια και να οριοθετηθεί. Πρώτο πρόβλημα αυτό. Δεύτερον, η εγγραφή δικαιωμάτων που είναι δικαιώματα ιδιοκτησίας προκαθορισμένα και σύμφωνα με τον νόμο. Γιατί ο νόμος λέει τη στη Μαδαγκασκάρη ότι ένα αγροτεμάχιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται επί 20 χρόνια, αλλά χρησιμοποιείται δεν σημαίνει ότι κατοικείται από κάποιον εδώ και γενιές, αλλά σημαίνει ότι θα πάρει την αξία του από τις αρχές που θα παρέμβουν όταν η Επιτροπή ζητήσει αυτό το τίτλο. Και τέλος, αν μπορέσει ο χωρικός αυτός να πάρει τον τίτλο στα χέρια του θα πρέπει να τον ενημερώνει κάθε φορά. Κάθε φορά που υπάρχει δηλαδή κάτι που γίνεται θα πρέπει να πηγαίνει να αλλάζει την εγγραφή στο κτηματολόγιο. Ποιο έχει τη δυνατότητα να το κάνει, ποιο έχει το χρόνο να το κάνει, ποιο ξέρει ότι πρέπει να το κάνει. Στη Μασκάρη υπάρχουν 29 υπηρεσίε ε, για το σύνολο. της επικράτειας. Δηλαδή 1200 χιλιόμετρα στη μία κατεύθυνση, 600 χιλιόμετρα στην άλλη κατεύθυνση είναι η χώρα αυτή και υπάρχουν μόνο 29 υπηρεσίες. Είναι λοιπόν αδύνατον οι χρήστες να φτάσουν στο σύστημα αυτό και λόγω του κόστους. Γιατί περίπου 500 δολάρια χρειάζεται για ένα χωρικό να πάρει ένα τίτλο κτηματολογίου σε μια συνήθεια αγροτεμάχιο 2-3 εκταρίων. Ποιος έχει τα χρήματα αυτά σε μια χώρα που μια οικογένεια δεν έχει ούτε ένα δολάριο την ημέρα. Το πρόβλημα δεν είναι στο τι γίνεται με το ΑΕΠ κλπ. Αλλά ότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί, ιδίω στην Ήπεθρο, είναι άτομα που ζουν συνεχώς σε αβεβαιότητα. Δεν πρόκειται για μια αβεβαιότητα του αλλά του εισοδήματο που θα τους επιτρέψει να επιζήσουν. Μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη με στα πλαίσια της πολιτικής ε, για τη γη. Αλλιώ δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό από το 2005 η Μαδαμασκάρη εισήγαγε ένα άλλο σύστημα, το λεγόμενο της ιδιοκτησίας gas. Είναι κάπως παρόμοιο αυτό που γίνεται στη Ρουάντα, στην Τανζανία και σε πολλές άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή στο επίπεδο των τοπικών αυτοδικήσεων, 1500 περίπου στην Δαμασκάρη, υπάρχουν, ε, υπάρχουν υπηρεσίες για τη γη που αποτελούνται θηρίδα γης που διαχειρίζονται την γεωιδιοκτησία σε τοπικό επίπεδο εφόσον δεν υπάρχουν τίτλοι κτηματολογίου. Τι τη χρηματολογία δίνονται μόνο από το κράτος, αλλά σας είπα αυτή είναι πολύ απομακρυσμένη από την πραγματικότητα. Σε τοπικό επίπεδο λοιπόν, εάν κάποιος θέλει να αποκτήσει τίτλους για την ιδιοκτησία του, θα πάει στην τόπια εκεί υπηρεσία που θα εισαγάγει μια επιτροπή αναγνώρισης των τοπικών δικαιωμάτων. Μια επιτροπή η οποία συνενώνει ε, κάποιους από την ε, υπηρεσία, τους επίσης του Ρεγιαμαντρίν που είναι η σοφή αν θέλετε, τόπια και επιτόπου και βέβαια όλους τους χρήστες, τους γείτονες που τους ενδιαφέρει η διαδικασία για να μπορεί αντιφατικά να γίνει καταγραφή. Τι γίνεται έτσι. Η διαδικασία αυτή, όπως είπε και η Άρα προηγουμένως, επιτρέπεται να επιληθούν επιτόπου, εκ των προτέρων πολλές φορές, πολλές από τις συντρούσεις. Στο σύνολο των ε, πιστοπτικών που έχουν δοθεί στη Μεταγασκάρη, το ποσοστό συγκρούσεων που διέκοψαν την διαδικασία δεν είναι ούτε καν 5% των αιτήσεων. και όλοι διακανονίστηκαν στους επόμενους δύο μήνες. Είμαστε λοιπόν σε ένα σύστημα που επιτρέπει να εξασφαλίσουμε αυτό που γίνεται. Θα σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Το αποτέλεσμα αυτών, και σας το λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κατανοήσουμε καλύτερα, 1.500 υπηρεσίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Θεωρητικά στην πράξη υπάρχουν 600 αυτές ε, τις θηρίδες ε, γης ε, στη Μαδανασκάρη, 29 υπηρεσίες κρατικές. Έξι υπογραφές χρειάζονται για τους τίτλους. Στη μία περίπτωση, στην άλλη κάθε δήμαρχος μπορεί να υπογράψει. Κόστος. Το πιο ακριβό, ακριβό σε τόπιο επίπεδο είναι το 10% και ούτε καν του δημόσιου τομέα. η διάρκεια επίσης υπάρχουν στο κράτος εκκρεμούσες αιτήσει από τη δεκαετία του 50. Από το 96 έχουν περίπου εγγυηθεί 500.000. Από το 2006 140.000 αιτήσει για τα πιστοποιητικά, 47 έχουν ήδη εγκριθεί. Ωραία είναι αυτά, αλλά δεν επιλύουν όλα τα προβλήματα. Και γιατί δεν επιλύουν όλα τα προβλήματα, γιατί έγινε ένα σφάλμα ώστε να φέρει μία από τις φιλοδοξίες της πολιτικής να εξασφαλιστεί η επένδυσή τους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα της επένδυσης. Αυτό που είναι τη κληρονομιά που θα δώσουν στα παιδιά τους. Το άλλο δεν του ενδιαφέρει. Ένα πρόβλημα αυτό. Δεύτερο πρόβλημα. Είχε προβλεφθεί μια που υπάρχουν ε, επενδύσεις και μικροπιστώσεις να βελτιωθεί η κατάσταση των εκμεταμοχείων στους οποίους υπάρχουν, για τα οποία υπάρχουν ε, πιστοποιητικά, αλλά δεν κάνουν τίποτα σχετικά οι χωρικοί. Το σύστημα λοιπόν από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται να επανεξεταστεί. Ίσως χρειάζεται και γι' αυτό είναι καλή συζήτηση σήμερα να σκεφτούμε αυτό που εμείς αποκαλούμε ε, ιδιωτική ιδιοκτησία. Τέλος, ο αριθμός των αγροτονοχείων και το μέγεθος ορισμένων από αυτά, όπως και σε άλλους χώρους που αναφέρθηκαν, υπάρχουν ε, αγροτομάχια που είναι 2 επί 3 μέτρα. Άμα χρησιμοποιήσετε το GPS για να το βρείτε, Θα έχετε αρνητικό αγροτεμάχιο, για να το πούμε έτσι ηρωνικά. Μπορείτε να το που, που... Βιάστηκα κύριε Πρόεδρε. Πολλά ξέχασα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά για την πιο τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση του τι γίνεται στην Μαδαγασκάρη. Ας μην ξεχνάμε τι προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν προσπαθούμε να καταγράψουμε μη καταγραμμένες γιές. Δεν θέλουμε να πάρουμε τους ελευθερόμενους από τις διοκτησίες ε, σε, σε σλάμ και να τους εγγράψουμε κάπου αλλού. Όχι, κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε κεφάλαιο Όλες οι καταγραφές που γίνονται και στη Ρουάντα που ακούσαμε, τα 8 εκατομμύρια αυτά αγροδομάχια που θα μπορέσουν να καταγραφούν στη Ρουάντα, όταν καταγραφούν γίνονται κεφάλαιο τμήμα μιας διαδικαθυσίας δημιουργίας πλούτου. Εγώ έχω ένα διαμέρισμα στο Σατολάν, αλλά δεν έχω, αν σας έλεγα ότι δεν έχω τίτλους γι' αυτό, δεν μπορώ να σας το πουλήσω, και μπορώ όμως να το κληρονομήσω στο γιο μου. Αν έχω τίτλους όμως μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να πάω στην τράπεζα να το καταθέσω τον τίτλο και πάνω σε αυτόν να δανειστώ χρήματα για να αγοράσω αυτοκίνητο ή άλλο, ή άλλο σπίτι ή κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να επανακεφαλοποιήσουμε για τις αναπτυσσόμενες χώρες το πλούτο αυτό. Και αν το κάνουμε αυτό, αν το πετύχουμε αυτό, σύμφωνα με τον νόμο της Σότο, θα δημιουργήσουμε 17 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε πια πολύ χρόνο. Έχουμε εδώ μια συζήτηση προβλέψει. Να κάνω μερικέ σκέψει. Καταγραφή. Το συζητήσαμε αυτό. Καταγραφή σε ένα βιβλίο ενώ Σε ένα κτηματολόγιο και να πάρει κανένα μια απόδειξη. Η καταγραφή τη γραφή στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλά θέματα σχετικά με αυτό που θα μπορούσαμε να συστήσουμε. Η Κομισιόν θα μπορούσε ίσως να μας κάνει μια παρουσίαση. Δεν θα ήθελα να καθυστερήσω τη συζήτηση, υπάρχουν πολλοί ομιλητές. Θα ήθελα απλώ να πω ότι ο λόγο που προωθούμε την πολιτική αυτή είναι μια πολιτική που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να απτυχθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πραγματικά να το λάβει αυτό υπόψη τη. Και να σα πω για ποιο λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί με την πολιτική για την κατοχή γη. Καταρχά, να σα πω ποια είναι η εμπειρία που έχουμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, τη χώρα που γνωρίζω καλύτερα, την Ιρλανδία. Μια εμπειρία την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Ο λόγος που έχουμε ένα διχασμένο νησί έχει να κάνει ακριβώ με την διοκτησία γης. Ένα μικρό τμήμα της γης δόθηκε σε ανθρώπους στην βόρειο-ανατολική Ιρλανδία, εργάστηκαν στην γη αυτή, χτίσανε σπίτια, επένδυσαν, κατάφεραν να δημιουργήσουν κεφάλαιο. Στο υπόλοιπο όμως του νησιού, στο υπόλοιπο της Ιρλανδίας, είχαμε κυρίως ε, αγροτεμάχια τα οποία ανήκανε σε ε, Βρετανούς οι οποίοι ε, ουσιαστικά εκμεταλλεύονταν πάρα πολλούς εργαζόμενους στα αγροτεμάχια αυτά που ήταν πάρα πολύ φτωχοί. Η Ιρλανδία μάλιστα είχε μεγαλύτερο πληθυσμό από την Αγγλία την εποχή εκείνη. Με την πάρθο του χρόνου λοιπόν τα πάντα περιστρέφονταν γύρω από την ε, ιδιοκτησία γης, γύρω από τη μίσθωση της γης. Και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα το ζήτημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της ε, δικής μου πολιτικής ζωής, είχαμε μια επιτροπή, την Land Commission, Επιτροπή για την Γη, για την Κατοχή Γης και είχαμε μάλιστα και έναν υπουργό αρμόδιο για την γη, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70. Δεν ξέρω αν είχαμε ακόμα και τη δεκαετία του 80 τον υπουργό αυτό. Θα έλεγα λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αξίζει να μελετήσει το μοντέλο αυτό, το πρότυπο αυτό. Αναφέρομαι σε μία χώρα η οποία αποτελούσε τμήμα μιας αυτοκρατορίας μια εποχή χώρα η οποία επλήγει αρκετά πρόσφατα και από την ένδια, την πείνα και το ζήτημα αυτό συνέβαλε πάρα πολύ στον τρό, στην εξέλιξη που είχε η χώρα αυτή. Αξίζει λοιπόν να μελετήσουμε το μοντέλο αυτό και αναφέρομαι σε μια εποχή πριν τους υπολογιστές, πριν την τεχνολογία που έχουμε σήμερα, πριν τους δορυφόρους. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία του Διαστήματος και θυμάμαι σε μια παρουσίαση που κάναν στο Στρασβούργο ότι ε, είπανε ότι μπορούσαν να δούνε από το δορυφόρο αν ένα αγροτεμάχιο βρισκόταν σε καθεστώς αγρανάπαυσης ή όχι. Και χρησιμοποιούν τους δορυφόρους αυτούς όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στη Σιρλάνκα, για παράδειγμα μετά το τζουνάμι, προκειμένου να καταφέρουν να εντοπίσουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και δώσανε συγκεκριμένες φωτογραφίες προκειμένου να δείξουν ποιο τμήμα της γης θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί, ποιο τμήμα της γης ανήκει σε ποιον και το καθεξής. Θεωρώ λοιπόν ότι θα μπορούσαμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που έχουμε ως κράτη-μέλη και την τεχνολογία που διαθέτουμε πλέον ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όταν πήγα στην Ρουάντα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το ότι έχουν πλέον ένα σύστημα κτηματολογίου, κάτι το αντίστοιχο τουλάχιστον με το κτηματολόγιο και υπάρχουν εκεί πέρα άτομα τα οποία έρχονται από την Βρετανική, την Ολλανδική υπηρεσία κτηματολογίου που βοηθούν τους εργαζόμενους στην Ρουάντα να στήσουν και τη δική τους υπηρεσία. Και βέβαια, συμβουλεύουν τους ανθρώπους εκεί στην Ρουάντα, δεν τους επιβάλλουν συγκεκριμένες πρακτικές, δεν τους λένε τι πρέπει να κάνουν. Στην Ρουάντα είδα ότι έρχονται σε επαφή πραγματικά με τους ανθρώπους, είναι σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών, οργανώνουν ακόμα και παιχνίδια ποδοσφαίρου με τον τοπικό πληθυσμό, προσπαθούν να έρθουν πιο κοντά στους ανθρώπους. Κατά αυτόν τον τρόπο οι πολίτες συμμετέχουν οι ίδιοι ενεργά και δεν θεωρώ ότι είναι εφάνταστο αυτό το οποίο λέμε. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω εγώ είναι ότι το μοντέλο το οποίο ακολουθήθηκε στην Ιρλανδία πραγματικά βοήθησε την εξέλιξη της ε, χώρας και στο Δουβλίνο, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, υπήρχαν πάρα πολλοί οικισμοί οι οποίοι δεν είχαν περάσει το κλιματολόγιο και στη συνέχεια τα αγροτεμάχια αυτά ιδιωτικοποιήθηκαν και πέρασαν στο κλιματολόγιο και εκδόθηκαν τίτλοι για τα αγροτεμάχια αυτά τα οποία δεν είχαν καταγραφεί στο παρελθόν. Και αυτό άλλαξε εντυπωσιακά τη ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι είχαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα κτήματα αυτά ω εγγύηση προκειμένου να έχουν μια οικονομική δραστηριότητα κερδοφόρα στη συνέχεια. Δεν μπορούν αυτά να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει, και αυτό θέλουμε να πετύχουμε άλλωστε μέσω της ακρόασης αυτής, να έχουμε μια νέα πολιτική διαχείρισης της γης, και νομίζω ότι όλε οι πολιτικέ ομάδε συμφωνούν με αυτό. Τουλάχιστον η σοσιαλιστική πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει, να ακολουθηθεί δηλαδή και το δικό μα παράδειγμα στι αναπτυσσόμενε χώρε, να χρησιμοποιήσουμε την συσσωρευμένη εμπειρία που έχουμε και δεχομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε στα πλαίσια τη αναπτυξιακή βοήθεια να προωθήσει περισσότερο τι προτεραιότητε αυτέ. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ του ομιλητές, πρόεδρο. Θα μπορούσα να ζητήσω από τον ε, Βιμ Άλτοφ να μας πει κάποια πράγματα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βιμ Άλτοφ ονομάζομαι, εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ασχολούμαστε με ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων. Σας ε, ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση της ακρόασης αυτής. Ευχαριστώ πολύ που φέρνετε πάλι στο προσκήνιο το σημαντικότατο αυτό ζήτημα. Ο κύριος ε, Μίτσελ πριν από λίγο είπε ότι α, όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να, γνωρίσουμε πόσο να αναγνωρίσουμε τις... πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα της γης. Με Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία του ζητήματος αυτού και θέλει να προωθήσει το ζήτημα περισσότερο μέσω των πολιτικών της. Είναι στις προτεραιότητές μας το ζήτημα αυτό και αυτό φαίνεται άλλωστε από την δημοσίευση των ε, κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μεταρρύθμιση της γης και για τη διαχείριση της γης, κατευθύντηρες γραμμές που δημοσιεύσαμε το 2004 και θεωρώ ότι το κείμενο αυτό παραμένει πολύ εύχριστο, ένα κείμενο πολύ σημαντικό, ένα κείμενο το οποίο μπορεί να δώσει καθοδήγηση. Στο έγγραφο αυτό, και σε αυτό αναφέρθηκαν άλλωστε και κάποιοι από τους ομιλητές δίνονται κάποια σημαντικά μηνύματα. Λέμε στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές ότι κάθε φορά που μιλάμε για γη δεν υπάρχει μία λύση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή από τον τοπικό πληθυσμό και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες και ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου οι διαδικασίες αυτές να λειτουργήσουν και να αποφέρουν αποτελέσματα. Το πιο σημαντικό όμως ε, ζήτημα είναι η ασφάλεια της πρόσβασης στη γη και η εξασφάλιση στην πρόσβαση σε δικαιώματα ιδιοκτησία. Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα του όλου ζητήματο κάθε φορά που μιλάμε για γη και σχετική πολιτική. Και επανέρχομαι στα εισαγωγικά σα σχόλια, κύριε Πρόεδρε, όταν ε, αναφερθήκατε στην αυξανόμενη ευημερία και στο αυξανόμενο εισόδημα και όταν είπατε ότι αυτά από μόνα τους δεν αρκούν, γιατί η ιδιοκτησία είναι κάτι το εξίσου σημαντικό. Μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ευμερία, την βάση για την πρόσβαση σε περαιτέρω πόρους. Μπορεί να αποτελέσει την, το χώρο παραγωγής πολλών σημαντικών προϊόντων. Όλα αυτά τα στοιχεία τα τονίζουμε στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τονίζουμε επίσης και το σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι οργανισμοί, οι διάφοροι φορείς, τα θεσμικά όργανα. Και αυτό φάνηκε άλλωστε και από τις παρουσιάσεις που γίνανε σήμερα το πρωί. Πόσο σημαντικό είναι να στήσουμε τα θεσμικά κοινά όργανα τα οποία θα βοηθήσουν στην στον κτηματογραφικό σχεδιασμό και στην καταγραφή και την καταχώρηση της γης. Επίσης, στις ε, κατευθυντήρες αυτές γραμμές Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέμε πώς θα πρέπει να γνωρίσουν πολλές φορές τα συστήματα που λειτουργούν βάσει θυμικού δικαίου. Δεν θα πρέπει αυτά να αποκλειστούν από την πολιτική την οποία ακολουθούμε, γιατί όπως σας είπα δεν υπάρχει μία μαγική λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν θέλουμε λοιπόν να αποκλείσουμε τις εθιμικές πρακτικές στις επαφές που έχουμε με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Από πιο πρακτικής πλευράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των προγραμμάτων των αναπτυξιακών προωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο διάφορα, διάφορες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις κατευθύνες γραμμές της ε, Αφρικανικής Ένωσης όσον αφορά την διοκτησία της γης, ε, κατευθύνες γραμμές που υποστηρίζει και το UN Habitat των Ηνωμένων Εθνών και σε χώρες όπως η Ρουάντα, το Μπαγκλαντές, στη Βενεζουέλα και στο Βιετνάμ έχουμε άμεση συμμετοχή. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα προγράμματα παγκοσμίω τα οποία εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζουμε. Προφανώς προσβλέπουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα όπου αυτό ενδείκνεται και όπου αυτό είναι δυνατό. Χωρί να ήθελα τώρα να προκαταβάλω τη συζήτηση που θα γίνει στο δεύτερο πάνελ, θα ήθελα να πω ότι ένα από τα ζητήματα που δεν καλύφθηκε αρκετά στι γραμμές γραμμέ Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ζήτημα των μεγάλων επενδύσεων μεγάλης κλίμακας που θα μπορούσαν να γίνουν στα πλαίσια των εθνικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή και των επενδύσεων αυτών που θα μπορούσαν να γίνουν σε μικρότερη κλίμακα όσον αφορά δηλαδή κάποια μικρά αγροτεμάχια και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ε, υπάρχουν άλλοι συναδελφοί μου όμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι σήμερα μαζί μου που θα μπορούσαν να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες ως προς αυτό. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, ο άλλο ομιλητή της Επιτροπής να συγκεντρώσει την προσοχή του στο, και να επικεντρωθεί στα δικαιώματα ιδιοκτησία. υπάρχει κάποιο άλλο από την Επιτροπή που θέλει να πάρει το λόγο. Uh, uh, Μήπω μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση, Πρόεδρε. Μάλιστα. Εάν θα πάρετε το λόγο, θέλετε κι εσεί να επικεντρώσετε στο θέμα μας που είναι δικαιώματα, ιδιοκτησία, χρηματολόγιο. Όχι στη γη μόνο από τη σκοπιά της αγροτικής γης, αλλά ε, και τη γη που δεν χρησιμοποιείται, για παράδειγμα. Ε, την, ε, την, την άγωνη γη, την ε, δικαιώματα ιδιοκτησίας γενικά. Το βασικό ζήτημα είναι ότι στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γη αναφερόμαστε στην αναγνώριση των, του εθνικού δικαίου όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας δεν λέμε ότι η καταχώρηση δεν είναι χρήσιμη. Ενδεχομένως χρειάζεται έτσι και αλλιώς. Αλλά η διαδικασία που οδηγεί στην καταχώρηση, στην εγγραφή σε πολλές χώρες, ίσως αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο που δεν λαμβάνει υπόψη τις αδυναμίες των θεσμών εμπροκειμένου, δηλαδή σε ενισόμενες χώρες. Καθώς επίσης και το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια όπου έχουμε την εντύπωση ότι μπορεί να αναπτυχθεί πιο γρήγορα ένα κτηματολόγιο. Για παράδειγμα, στις χώρες όπως η Ρουάντα, όπου ασκείται πίεση σε επίπεδο πληθυσμού και η ανάγκη για καταχώρηση γίνεται πιο αισθητή από ό,τι σε χώρες όπου δεν υπάρχει αυτή ε, η πίεση, ε, η ανάπτυξη του πληθυσμού, η, το πρόβλημα με τους, με τους πόρους ε, και κάτι άλλο. Στις αναπτυσσόμενες αστικές περιοχές, εκεί, εκεί είναι πιο επίγουσα η ανάγκη για την ύπαρξη αυτών των συστημάτων καταχώρησης. Ευχαριστούμε. Αν λοιπόν και εσείς το αναγνωρίζετε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής γης θα μπορούσαμε να τα βάλουμε ε, και στα ε, στρατηγικά μας έγγραφα. Όταν λοιπόν εξετάζουμε ε, την πρόοδο, τότε το όχι μόνο το νερό, αλλά και η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην υγεία, αλλά και τα δικαιώματα ιδιοκτησία θα μπορούσαν να είναι εξίσου σημαντικά. Να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους του Κοινοβούλιο. Θέλετε να πείτε κάτι. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Ντίβα που μου δίνετε το λόγο και που διοργανώσετε αυτή τη συζήτηση. Παρόλο που εγώ θα πρέπει να εκφράσω μία αντίθετη άποψη ή προκλητική. Είπατε ότι το θέμα είναι δημιουργία κεφαλαίου και πλούτου. Το θέμα είναι για ποιον και αυτό για μένα είναι το βασικό ζήτημα. Πολλοί οικονομολόγοι και πολιτικοί ε, τον συγχρονισμό, την ανάπτυξη, ε, το ταυτίζουν με την ε, ατομική ιδιοκτησία. Αλλά εγώ δεν είμαι πεπισμένη για το ότι η ιδιωτικοποίηση της γης και η κατανομή τους σε ιδιωτικό επίπεδο είναι, το, είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές η γη είναι κοινό αγαθό και πολλές φορές ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο. Πρόσφατα, το 2007, ε, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ε, υιοθέτησε μία διακήρυξη για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών, ε, όπου συμπεριλαμβάνει μία ρήτρα που αναφέρει το εξή. Οι αυτόχθονοι λαοί έχουν το δικαίωμα στη γη, ε, στη γη, ε, στο έδαφος και στους πόρους που, ε, εκεί όπου κατοικούν κατά παραδοσιακό τρόπο που χρησιμοποιούν ή που απέκτησαν. Και πρόσφατα και εγώ υπέβαλα μια τροπολογία που, που έγινε δεχτή από το Κοινοβούλιο εν ώψη του ψηφίσματος για τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα στην Κοπεχάγη. Εκεί πάλι μιλούσαμε για τους αυτόχθονες και τους ενδογενείς και αναγνωρίζαμε το δικαίωμά τους στη συλλογική ιδιοκτησία των αυτόνομων ανδογενών περιοχών. Ε, ρωτώ λοιπόν, πώς βλέπετε να συνδέεται το θημικό δίκαιο το τα αναγνωρισμένα δικαιώματα ε, των αυτοχθόνων ε, ε, στη γη τους και την ιδιωτικοποίηση που ορισμένοι θεωρούν ότι είναι το μοναδικό εργαλείο για την ανάπτυξη. Και αν επιτρέπετε, να σας πω το εξή. Ξέρω ότι τώρα μιλάμε για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά αυτή η συζήτηση μου θυμίζει ένα αριθμό το οποίο, τον οποίο δεν μπορώ, να το ξεχάσω. Κάθε τρία λεπτά ε, κλείνει μια γεωργική εκμετάλλευση εδώ στην Ευρώπη. Και κάποιος άλλος αναφέρθηκε ε, στο πραγματικό πρόβλημα. Η πρόσβαση στη γη και κοιτάξτε, βλέποντα το πόσο κλείνουν οι γεωργικέ επιχειρήσει, πόσε γεωργικέ επιχειρήσει κλείνουν στην Ευρώπη, ε, τελικά δεν στερούμε από του νέου το δικαίωμα στην πρόσβαση στη γη. Γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με, τη βιωτική, με την ατομική ιδιοκτησία, την υπερχρέωση κτλ. Θα ήθελα λοιπόν αυτή η συζήτηση, είτε εδώ είτε σε ανεψόμενε χώρε, να μην ε, συνδέεται, να συνδεθεί και με το ε, εξή ερώτημα. Πώ θα γίνει η πρόσβαση στη γη, πώ θα εγκατασταθούν οι νέοι ε, σε αγροτικέ περιοχέ. Και αυτό ανεξάρτητα από τη σύνδεσή του με την ιδιοκτησία. Αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι η εγγύηση του δικαιώματο τη πρόσβαση στη γη και όχι απαραίτητα ε, συνδέοντάς το με την ατομική ιδιοκτησία της γης. Finally, Επιτέλους, μια πολιτική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσαν ε, οι ομιλητές να απαντήσουν. Κλέιτον, Λαρίσα. I, think on some level... Κοιτάξτε, αυτή η διάκριση ανάμεσα στη συλλογή και στην, ε, ιδιωτική, και στην τομική ιδιοκτησία ε, κατά κάποιο τρόπο μας ε, ε, κάνει να ξεχνάμε το βασικό πρόβλημα. Μπορεί... Ε, κοίταξε, έχουμε δύο ανθρώπου που μένουν στο ίδιο σπίτι. Δύο ανθρώπου ε, που εργάζονται πάνω στο και την ίδια γη. Άρα εκ των πραγμάτων έχουμε μία ε, συμβίωση, αν θέλετε, μία συλλογική χρησιμοποίηση και αξιοποίηση. Το πρόβλημα εδώ όμω είναι το εξή. Και το πρόβλημα που αναφέρατε έχει να κάνει με την εγγύηση του δικαιώματο πρόσβαση στη γη. Και φοβάμαι ότι δεν καταλάβατε αυτό που θέλω να πω στην ομιλία μου είναι η διαχείριση του ανταγωνισμού. Έχουμε δηλαδή ε, ε πόρου που θέλουν όλοι να του καταλάβουν ταυτόχρονα. Πώ λοιπόν μπορούμε να αξιοποιήσουμε ε, ε, το πρόβλημα αυτό έτσι ώστε να υπάρχει ε, αγορά ε, φθηνών πόρων και μετατροπή του σε πλούσιου πόρου. Όταν μιλούμε για του ενδογενού πληθυσμού, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η κοινότητα ω τοπική κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ ότι ερχόμαστε και τα βλέπουμε τα πράγματα κάτω από την εξουσία του κράτου. Αγνοούμε το γεγονό ότι κατά παράδοση ενδογενή κοινότητα έχουν προνόμια όσον αφορά την, ε, τη συμπεριφορά του και τη ζωή του. Συμφωνώ σίγουρα ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μα στο ζήτημα αυτό. Σε πολλέ χώρε όπου γίνεται παραβίαση αυτών των παραδοσιακών δικαιωμάτων. Αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις η συλλογική ιδιοκτησία εκ μέρους μιας κοινότητας και αυτή η αντίσταση στην έννοια της ιδιωτικοποίησης είναι κάτι το ιδεολογικό. Με την έννοια ότι σε αυτές τις περιπτώσεις Υπάρχει ατομική ιδιοκτησία μέσα στις κοινότητε σε οικογενειακή βάση. Αν πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι η ιδιοκτησία της κοινότητα, με αδιέρετο τρόπο, αλλά η κοινότητα μπορεί να είναι κάτι τόσο Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε ποιο απαρτίζει την κοινότητα, ποιο έχει αυτά τα δικαιώματα συγκεκριμένα. Και στην ουσία καταλήγουμε στην ίδια διαδικασία. Να είναι τα πάντα ορατά και ρητά, να μην υπάρχει καμία ασάφεια που να οδηγεί σε συγκρούσει. Ε, ε, ε, δηλαδή ασάφεια λόγω ασαφών κανόνων. Πριν δώσω το λόγο στην Κλαρίσα, να, να ρωτήσω την Άννα, τι είδατε επί τόπου στη Ρουάντα όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Αν κατάλαβα καλά, υπάρχει ένα πρόβλημα με την ιδιωτική ιδιοκτησία ως τη λύση, ως την πανάκια. Και εδώ θέσατε το, βασικό ερώτημα από τη σκοπιά της προ... του δικαιώματο πρόσβαση στη γη. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχει συζητηθεί ευρέω στη Ρουάντα το ζήτημα αυτό. Η ατομική ιδιοκτησία θεωρείται ω κάτι το δεδομένο. Η Μοζαμβίκη είναι πιο ενδιαφέρον παράδειγμα. I mean, is... Γιατί εκεί όχι μόνο ε, η γη, το κράτος ε, είναι ιδιοκτήτης ολόκληρης ε, της γης που μισθώνει τη γη στη συνέχεια, αλλά δεν επιτρέπονται και οι συναλλαγές και οι αγοραπολισίες. Εκεί λοιπόν γίνεται συζήτηση και προβληματισμό σε, ευραίο, σε ευρύ επίπεδο, σε ευρύτερο επίπεδο, για το κατά πόσο πρέπει να επιτρέπονται αυτές οι συναλλαγές επίπεδο γης. Στη Μοζαμβίκη, Υπάρχει και αναγνώριση από τον νόμο της κοινοτικής ιδιοκτησίας. αν κανείς ε, ε, ε, αξιοποιεί τη γη για 10 χρόνια ή ανήκει ε, σε μία κοινότητα, θεωρείται ότι, ότι θεωρείται ότι μπορεί να χρησιμοποιεί την, τη γη αυτή. Δηλαδή δεν, είναι, δεν είσαι ιδιοκτήτης, αλλά έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιείς τη γη. Καταλαβαίνω ότι το μιλάτε για πρόσβαση δεν εννοείται τη φυσική πρόσβαση, αλλά εννοείται την αξιοποίηση. Λοιπόν, κοιτάξτε. Κοιτάτε κάποιον που 29 ο είχε 14.000 ε, acres και μετά το υπόλοιπο ε, μου το πήρανε και το ε, δώσανε σε εκείνους που καλλιεργούσαν τη γη. Αυτοί οι άνθρωποι γίνανε πλούσιοι αν θέλετε ε, και μπόρεσαν έτσι να χρησιμοποιούν σουν τη γη. Ε, κοιτάξτε. Υπάρχει κάποιος που λέγεται Pat the Cope Kalahar. Είναι ότι πάρα πολλοί Kalahar υπάρχουν στο Ντόνεγκαλ και ο παππούς του ήταν εκείνος που είχε μια ε, um, ένα συνεταιρισμό. Λοιπόν, υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα όταν υπάρχουν αυτόχθονοι πληθυσμοί κλπ. Εγώ δεν ξέρω, γιατί εμείς κάνουμε κάτι για τους εαυτούς μας και ελέγχουμε τους όρους που δεν κάνουν το ίδιο. Στην Ελλάδα, παραδείγματος, όταν άρχισε να υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, δεν άλλαξαν όλοι ε, την πολιτική τους. Εμείς δεν έχουμε και πολύ συντηρητική παράδοση στην Ιρλανδία, αλλά τι έγινε. Άλλαξε η μακροπρόθεσμη επένδυση των ε, πολιτών στην κοινότητά τους. Όταν εγώ πάω στη Ρουάντα στην Αγγόλα και βλέπω όλους αυτούς που έχουν τα κινητά και ξέρω ότι είναι ευφυείς άνθρωποι με φιλοδοξίες. Όπω έπεσε το τείχο του Βερολίνου, έτσι και το τείχο του Βερολίνου τη φτώχεια στην αναπτυσσόμενη χώρα κάποια στιγμή θα πέσει. Μα είναι το ίδιο όπως εμείς και έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες που έχουμε εμείς. Θέλουν να έχουν λίγη γη, να επενδύσουν, να δώσουν κάτι στα παιδιά τους. Γιατί αυτό που θεωρώ εγώ φυσιολογικό για μένα να μην το θεωρώ φυσιολογικό για τους άλλους. Μα εγώ ακριβώς το αντίθετο είχα πει κύριε Μίτσελ, ότι στη δική μας ε, κοινωνία, στη Γαλλία μιλάω, όχι σε άλλους, βλέπω 3 εκατομμύρια 700.000 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις ε, γης τους γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν τα δάνεια πάνω σε αυτή την ιδιοκτική ε, ιδιοκτησία. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να δώσουμε σε πολλούς ε, νέους γεωργούς να εγκαταστηθούν στη γη αυτή χωρίς να είναι ιδιοκτήτες και να μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν. Α, δηλαδή αυτό χτίζει ξανά όμως το τείχος του Βερολίνου. Αυτή η ιδέα εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Έχουμε κι άλλο ένα πάνελ. Ναι, αλλά ξέρω ότι ίσως ο Τσάρλς ξέρει να, υποβάλει κάποια ερώτηση. Τσάρλς Κόρεντς, θέλετε να υποβάλλετε μια ερώτηση. Όχι. Όχι. Ωραία. Ωραία. Κάποιος από το πάνελ που θέλει να απαντήσει, παρακαλώ. Κλάρισα. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση επί τόπου. Αφενός ε, την ε, τροποποίηση των υγειών και τον κοινωνικό παράγοντα που παίζει εδώ ένα ρόλο. Δεν ξέρω όμως σε ποιο επίπεδο γίνεται αυτό. έχουμε την κλίμακα, αν θέλετε, της ιδιοκτησίας. Μπορεί κανείς να ξεκινήσει από κάπου και να ανεβεί και να φτάσει σε δικαιώματα ελεύθερης χρήσης. Μπορούν να υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες εδώ μεταξύ. Ο καθένας πρέπει δηλαδή να ενταχθεί κάπου σε αυτή την κλίμακα, αν θέλετε. Και αυτό φαίνεται γίνεται επιτόπου για πρακτικούς λόγους και αυτό που βλέπουμε και μολόδα για τις αστικές περιοχές είναι ότι έχουμε ανεπίσημη ιδιοκτησία και επίσημη ιδιοκτησία και η αγορά της γης και της κατοικίας ε, λειτουργεί και για τις επίσημες και για τις ανεπίσημες. Θα ήθελα λοιπόν να πω και το ξέρω κύριο Μπλοκ ότι οι κατευθυντές που έχει προετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλές, αλλά δεν είναι έτσι συγκεκριμένες για τις αστικές περιοχές. Ίσως κάτι θα μπορούσαμε να μάθουμε από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι αγορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προέδρο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για, την, ε, για το τμήμα αυτό τη συνεδρίασης. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου Γκέι Μίτσελ τώρα να προεδρεύσει το υπόλοιπο. We need okay. to um, ask the panel to Πρέπει να παρακαλούσουμε το πάνελ να περάσει την πρώτη γραμμή να κάτσει και να έρθει το καινούριο πάνελ να κάτσει εδώ. Okay, while, while the panel is joining us, we, we only have about an hour left. Um, Κοιτάξτε, έχουμε μόνο μια ώρα ακόμα για το καινούριο πάνελ. Θα έλεγα, οι νέοι ομιλητές θα μιλήσουμε 10 λεπτά και να έχουμε μετά την ευκαιρία να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Okay, you're, you're all very welcome. I'm just going to keep moving if you don't mind because we, we're going to finish at 6, 6 o'clock. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 6. Σας ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο πάνελ θα ασχοληθεί με το ζήτημα της αρπαγής της γης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Φαινόμενο το οποίο επεκτείνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και θέλουμε να δούμε στα πλαίσια του πάνελ ποια μέτρα έχουν εγκριθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Το δεύτερο πάνελ αποτελείται από τέσσερις ομιλητές Roman Hair από το δίκτυο ανάληψης δράσης Food First την Βιολέτ Ρουπανέρ από το δίκτυο 3D της Γενέβης, το Michael Taylor, ο οποίος είναι program manager για το για το συνασπισμό παγκόσμιας πολιτικής ε, για την Αφρική και από τον Χένρι Σαραγκίκ που είναι γενικός στενιστής του οργανισμού Λαβία Καμπεσίνα της Ινδονησίας. Το λόγο έχει πρώτος ο Ρόμαν Χέρ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στα 10 λεπτά. Βλέπετε την παρουσίαση. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή ε, ε, μάλλον την Επιτροπή μας εδώ που κατάφερε να συνδυάσει τα δύο αυτά ζητήματα, το ζήτημα της ιδιοκτησίας με το ζήτημα της αρπαγής της γης. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται ο συσχετισμός αυτός και θα ήθελα να κάνω κάποια πρώτα σχόλια για το ζήτημα αυτό, να κάνω κάποιες δηλώσεις όσον αφορά το ζήτημα της αρπαγής της γης. Αν περιμένετε όμως να σας κάνω ένα κατάλογο συγκεκριμένων περιπτώσεων και συγκεκριμένων λύσεων θα σε απογοητεύσω. Καταρχάς, θα πρέπει να διευρύνουμε λίγο το φάσμα της συζήτησης. Εφόσον μιλάμε για την αγορά της γης, αναφερόμαστε πολύ συχνά μόνο στα πλαίσια της αγροτικής αλλά θα πρέπει να δούμε ότι μιλάμε πάρα πολλές φορές και για άλλε εκτάσεις που έχουν διαφορετικές ε, χρήσεις, όπως για παράδειγμα για τον τουρισμό, για την εξόριξη μεταλλευμάτων ή και εκτάσεις που καλύπτονται από δάση. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ τώρα στα αγροτεμάχια εκείνα που χρησιμοποιούνται κυρίω για γεωργικέ δραστηριότητε και να δούμε ποια είναι τα φαινόμενα αρπαγής γης για τα αγροτεμάχια αυτά να σας δώσω κάποια βασικά στοιχεία εκτιμήσεις της ΦΑΟ. Τα τελευταία τρία χρόνια μόνο και μόνο στην Αφρική 20 εκατομμύρια εκτάρια γης έχουν αποκτηθεί από ξένους επενδυτές. Άλλες εκτιμήσεις μιλάνε για 50 εκατομμύρια εκτάρια. Θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε μεταξύ τους τους αριθμούς αυτούς και πρέπει να σας πω ότι 100 εκατομμύρια εκτάρια είναι η συνολική καλλιεργήσιμη γη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, απόκτηση αυτή γης ε, ουσιαστικά έχει να κάνει με πολύ, χρονή μίσθωση που καλύπτει μια περίοδο 30 μέχρι 99 ετών. Σε ποιο πλαίσιο τώρα γίνεται το φαινόμενο αυτό της απόκτησης της γης. Το πρώτο σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω και το οποίο έχει να κάνει και με τη συζήτηση που κάναμε στο πρώτο πάνελ είναι το πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς της γης από τα μέσα της δεκαετίας του 90 η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι οργανισμοί πίεζαν πάρα πολύ για την ιδιωτικοποίηση και την απελευθέρωση της γης, δηλαδή να γίνει η γη διαθέσιμη για τους ξένους επενδυτές και για διεθνείς επενδυτές. Έχουμε επίσης το Millennium Challenge Account που είναι ένα διεθνές δίκτυο, αλλά έχουμε και κάποια επιμέρους δίκτυα εθνικά τα οποία προωθούν τέτοιες πολιτικές, επένδυσης δηλαδή σε γη στο εξωτερικό και πρέπει επίσης να σας πω ότι υπήρχε και μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στα αγροτεμάχια αυτά. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που έχουμε μας δείχνουν ότι στις αρχές δεκαετίας του 90 Περίπου ένα δισεκατομμύριο αμερικανικά δολάρια έχουν επενδυθεί σε αγροτεμάχια που προορίζονται για γεωργική εκμετάλλευση και το 2007 φτάσαμε τα 3 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Βλέπω τρεις βασικούς λόγους που οδηγούν σε αυτή την μεγάλη διαδικασία αλλαγής της ε, διάρθρωσης εκμετάλλευση της γης. Καταρχά έχουμε την κρίση όσον αφορά την τιμή των τροφίμων το 2008. Το ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων επανήλθε στις βασικές προτεραιότητες πολλών κρατών μελών και υπάρχουν πολλές πλούσιες χώρες στον κόσμο που από αποκαλείται ως offshore farming, προσπαθούν ουσιαστικά μέσω της δραστηριότητας που έχουν σε τρίτες χώρες να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό της χώρας σε τρόφιμα. Ο δεύτερος σημαντικός λόγος που οδηγεί στη μεγάλη αυτή ε, μεταρρύθμιση όσον αφορά τη χρήση της γης έχει να κάνει με τα καύσιμα τα οποία προέρχονται από αγροτικά προϊόντα. Υπάρχουν ε, όλο και περισσότερα αγροτικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καυσίμων. Έχουμε συγκεκριμένες ποσοστώσεις μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπεται ότι ένα 37% όλων των περιπτώσεων αρπαγής γης γίνεται ακριβώς για να παραχθούν αυτά τα βιοκάψιμα, καύσιμα τα οποία προέρχονται από αγροτικά προϊόντα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η συμβολή αν θέλετε των καυσίμων αυτών, πως ε, η παραγωγή των καυσίμων αυτών οδηγεί σε ε, ε, πολύ έντονα φαινόμενα αρπαγής γης. Βλέπουμε επίσης ότι περίπου 500 εκατομμύρια εκτάρια θα χρησιμοποιηθούν μέχρι το 2045 προκειμένου να έχουμε ένα βιώσιμο καθεστώς καυσίμων, προκειμένου να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε μια υφόρο ανάπτυξη στα γεωργικά καύσιμα. Επίσης έχουμε και τη γενικότερη οικονομική κρίση που συμβάλλει και αυτή ο σημαντικός ε, λόγος, ο σημαντικός παράγοντας. Υπάρχει μια γενικότερη μεγάλη αναζήτηση για πραγματικές νέες επενδύσεις επιτόπου σε διάφορες συναπτυσσόμενες χώρες από διάφορα, διάφορους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά ταμεία. Υπάρχουν τώρα βέβαια κάποια νέα φαινόμενα. Τι έχει αλλάξει στην όλη κατάσταση. Ένας χωρικός από την Καμπότζη ρώτησε πριν από λίγο γιατί αγοράζουν ουσιαστικά το σύνολο των γεωργικών μας εκτάσεων αντί να αγοράσουν τελικά τα προϊόντα μας, το ρύζι δηλαδή το οποίο παράγουμε εμείς στις περιοχές αυτές, στα αγροτεμάχια αυτά. Η Παγκόσμια Τράπεζα στο παρελθόν επένδυε περισσότερο σε γεωργικά προϊόντα, ενώ τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες επενδύσεις στα βιοκάψιμα. Επίσης επικεντρώνονται πλέον οι διεθνείς οργανισμοί στα, στις παραγωγές υψηλής αξίας, στα αγροτικά αυτά προϊόντα τα οποία παρέχουν υψηλή αξία, ιδίως αυτά που οδηγούν στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Επίσης ε, στην ε, Κεντρική Αμερική Ήδη από τη δεκαετία του 70 είχαμε κάποιες εταιρείες όπως η ε, Τσικίτα που εκμεταλλεύονταν 20 έως 50 εκατομμύρια εκτάρια. Τώρα έχουμε αντίστοιχες πολυεθνικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται παγκοσμίως εκατοντάδες εκατομμύρια καλλιεργήσιμης γης. Επίσης έχουμε και διαφορετικούς πλέον παράγοντες στα πλαίσια της αγοράς αυτής. Δεν έχουμε μόνο τον ιδιωτικό τομέα που δραστηριοποιείται πάρα πολύ, αλλά έχουμε και πραγματικές ε, χώρες. Έχουμε τον κρατικό κλάδο που άμεσα ή έμεσα επενδύει σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και βέβαια έχουμε και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη δράση. Πριν από ένα μήνα πήγα στην Καμπότζη και εκεί μαζί με συναδέλφους μου έκανα μία διερευνητική επίσκεψη και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις παρατηρήσεις μας, σε κάποια από τα πορίσματα της έρευνάς μας. Αν δείτε το χάρτη αυτό θα συνειδητοποιήσετε ότι με τα χρωματιστά αυτά σημεία στον χάρτη βλέπετε τις περιοχές εκείνες που έχουν εκχωρηθεί στο κράτος και βλέπετε ότι υπάρχουν μόνο κάποιοι πολύ μικροί διάδρομοι, κάποιες πολλές στενές και μικρές περιοχές που έχουν απομείνει τελικά για τους χωρικούς. Βλέπετε εδώ πέρα σε αυτή τη φωτογραφία την αποψήλωση ενός δάσους που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το τοπικό πληθυσμό. Στο δάσος αυτό ο τοπικός πληθυσμός προχωρούσε με την εκτροφή βουβαλιών και επίσης καλλιεργούσε διάφορα φρούτα, διάφορα δέντρα. Βλέπετε επίσης στην φωτογραφία αυτή πως έχει καταλήξει μία μικρή αλλιευτική κοινότητα βλέπετε ότι έχουν καταφέρει να καταχωρήσουν στα πλαίσια της θάλασσας αυτής που μάζει πλέον με ποταμό συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες τουλάχιστον μπορούν να συνεχίζουν με την ελευτική τους δραστηριότητα. Δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος της θάλασσας αυτής δεν τους παρέχεται πλέον για λήψη ακριβώς επειδή δεν τους ανήκει επίσημα, δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Πολλές φορές τις εξελίξεις αυτές όπως αυτές που σας περιέγραψα στην Καμπότζη τις έχουμε ή μάλλον γίνονται στο όνομα της ανάπτυξης και υπάρχουν και πάρα πολλοί εμπεδιτές που πηγαίνουν στη χώρα αυτή και υπόσχονται νέες θέσεις εργασίας, υπόσχονται τη δημιουργία υποδομών και υπόσχονται ανάπτυξη η οποία θα είναι υποφελής για όλους. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, οι ελάχιστες που δημιουργούνται παρέχουν πολύ χαμηλού μισθού, χαμηλότερου από αυτού που είχαν χωρικοί στο παρελθόν με τη δικιά του αγροτική δραστηριότητα και τι περισσότερε φορέ πρόκειται για καθαρά επισφαλή εποχιακή δουλειά και όχι για μόνιμε θέσει εργασία. Επίσης, η υποδομή που δημιουργείται όταν δημιουργείται δεν είναι για τον τοπικό πληθυσμό, αλλά προορίζεται περισσότερο για τις εξαγωγές, πρόκειται ουσιαστικά για λιμένες, για αυτοκινητοδρόμους. Όλα αυτά δεν βοηθούν τον τοπικό πληθυσμό, δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές και επίσης ε, χάνεται η πρόσβαση του τοπικού πληθυσμού σε δάση, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και σε θάλασσες υποταμούς που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν για την αλία. Επίσης, η πρακτική αυτή της αρπαγής της γης παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στην τροφή, επίσης αυξάνει την συγκέντρωση της ιδιοκτησίας της γης σε συγκεκριμένους ανθρώπους και εταιρείε και επίσης περιθωριοποιεί όλο και περισσότερο τους τοπικούς γηγενείς πληθυσμούς. Το ζήτημα λοιπόν αυτό παραμένει από τις βασικές μας προτεραιότητες και θεωρούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τις σωστές πρακτικές και όχι την ε, αναδιάρθρωση της αγροτικής γης που μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενέστερη θέση τους τοπικούς πληθυσμούς. Θεωρούμε επίσης ότι δεν θα πρέπει η επένδυση αυτή που γίνεται στις αμπτυσσόμενες χώρες να οδηγήσει σε βιομηχανική εντατική καλλιέργεια καταργώντας την τοπική καλλιέργεια που γινόταν από τους τοπικούς πληθυσμούς, μια καλλιέργεια βέβαια σε μικρότερη κλίμακα. Μπορώ να σας δώσω αντίστοιχα παραδείγματα και για άλλες χώρες πέρα από την Καμπότζη, όπως για την Κένια. Στην τελευταία αυτή διαφάνεια βλέπετε κάποιες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με κοινέ δράσεις που έχουν αναλάβει διάφοροι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη. Οι οργανισμοί αυτοί προσπαθούν να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόθεση της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως στην Αφρική. Επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο ζήτημα της αρπαγής της γης και σχετικές δραστηριότητες, πώς γίνεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από επιμέρους κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να κάνω μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δραστηριότητες τους που οδηγούν σε αρπαγή γης. Καταρχάς θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας διεθνής κανονισμός που να αποτρέπει το φαινόμενο αυτό της αρπαγής της γης, να έχουμε ένα νέο, πλέο επενδύσεων, ένα νέο πλαίσιο επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επενδύσεις στις τρίτες χώρες, όπου θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε ρήτρε για την μη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νέους κανονισμούς όσον αφορά τα βιοκαύσιμα και τα καύσιμα τα οποία παράγονται από αγροτικά προϊόντα, Επίσης, ε, νέες κατευθυντήρε γραμμές όσον αφορά την πρόθεση των ανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ε, τρίτες αναπτυσσόμενε χώρες και να γίνεται και μια νέα αναφορά όσον αφορά, ε, μια νέα φορά όσον αφορά την καλλιέργεια των ζωοτροφών στις χώρες αυτές, ζήτημα το οποίο προωθεί πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίση να σας πω ότι η δική μα οργάνωση προωθεί τι πρωτοβουλίες της Αφρικανικής Ένωση και αντίστοιχη προσέγγιση θα πρέπει να έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει τέλος να ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τις ε, εθελούσες κατευθυντήρες γραμμές ε, του ΦΑΟ όσον αφορά την κατοχή γης στις αναπτυσσόμενες χώρες και να συμμορφωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της με τα συμπεράσματα της ε, διάσκεψης, της παγκόσμιας διάσκεψης που έγινε πριν από λίγο καιρό όσον αφορά τη γεωργική μεταρρύθμιση και την άπτυξη της υπαίθρου, της διάσκεψης Κάρτε Ολοκληρώνω με το άρθρο 1 1-2 της ε, Διεθνούς Σύμβασης για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, άρθρο το οποίο έχουν ε, υπογράψει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύμβαση αυτή λέγεται ότι σε καμία περίπτωση οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να στερούνται από τα βασικά μέσα επιβίωσής τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση. Δεν ξέρω αν η γραμματεία θα μας μοιράσει αυτά τα έγγραφα που μας παρουσίασε. Το επόμενος ομιλητής είναι η Violet Τρούπενερ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ε, έρθω εδώ σήμερα και να σας δώσω τη θέση μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ και τους δύο πρόεδρους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω δύο λόγια για το 3D είμαστε. Είμαστε μια μη επικερδής οργάνωση στη Γενέβη με αποστολή την της ότιμης ε, οικονομίας ε, και ανάπτυξης όπου ε, όλοι να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα εγείρουμε ε, την, ε, ε, την προσοχή όλων όσων διαμορφώνουν την πολιτική στα ανθρώπινα δικαιώματα, σε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο κοινό κτλ. Και προσπαθούμε να το πράξουμε τονίζοντας το πώς συνδέεται η διεθνής πολιτική και η επίπτωση στα ανθρώπινα δικαιώματα επί τόπου. Το θέμα μου σήμερα, αφού ακούσαμε από, τον προηγούμενο μιλητή, για τους προηγούμενους για τις πραγματικότητες ε, ε, που αφορούν το ζήτημα της απόκτησης γης είναι να σας δώσουμε μια προοπτική ε, ανθρώπινα δικαιώματα και ε, το πώς μπορεί να βοηθήσει, με τι προσθέμενη αξία μπορεί να προσδώσει ε, η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ζήτημα αυτό. Τέλος, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, την υπεύθυνη επένδυση στη γεωργία και την πρόθεση του ζητήματος αυτού στα διεθνή φόρα. Σύμφωνα με τον ειδικό εισηγητή των για το δικαίωμα στην τροφή, σήμερα η κατάσταση οφείλεται αυτές τις προηγούμενες αποτυχίες. Ε, δήλωσε λοιπόν ότι αποτύχαμε στο, στο παρελθόν να επενδύσουμε παρκώς στη γεωργία και στην ανάπτυξη πέθρου. Αποτύχαμε να προωθήσουμε μέσα γεωργικής παραγωγής ε, που δεν καταστρέφουν το έδαφος ε, και δεν εξαντλούν τις υπόγει, τους υπόγειους σπόρους. και σήμερα αποτυγχάνουμε να θεσπίσουμε παγκόσμιες αγορές που να λειτουργούν σωστά και να είναι πιο αξιόπιστες, παγκόσμιες αγορές για τα γεωργικά προϊόντα. Ποια είναι λοιπόν, η, τι θα επιφέρει η προσέγγιση ανθρώπινα δικαιώματα στο ζήτημα αυτό. Πρώτα απ' όλα, όλα τα κράτη έχουν κυρώσει ε, τουλάχιστον μία από τις, ε, μία ε, από τις υφιστάμενες συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα λοιπόν σε θεωρητική βάση δέχονται να ε, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προβλέπονται οι μηχανισμοί για την ανάληψη ευθύνη και τη λογοδοσία. Και δεν μιλάμε εδώ για τη λογοδοσία σε επίπεδο κυβέρνηση, αλλά και σε επίπεδο οικονομικών εταίρων. Ε, και μπορούν ε, να ασκήσουν προσφυγή ε, είτε ομάδες είτε άτομα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν και τα τεκτενόμενα εντός των χωρών αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των χωρών και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν έτσι ώστε η δράση ή η αδράνεια δεν υπονομεύει τα δικαιώματα των πολιτών τους. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η υποχρέωση ρύθμισης της συμπεριφοράς των μη κρατικών εταίρων, για παράδειγμα των πολυεθνικών εταιριών. Τέλος, μια προσέγγιση ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ουδέτερη. Δεν ε, προασπίζεται ένα συγκεκριμένο είδο κυβέρνηση, ε, διακυβέρνηση πολιτικού συστήματος και δεν δίνει πολιτικές προδιαγραφές για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Δεν μιλά για συγκεκριμένα μοντέλα. Η βασική ιδέα είναι ότι αν μια πολιτική επιδρά αρνητικά στα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε ε, απαιτείται δράση από την ελόγω για την επανόρθωση της κατάστασης. Κανείς δεν υποστηρίζει ότι η επένδυση στη Γεωργία ε, είναι ανώφελη. Ε, το θέμα αυτό αφορά όλες ε, τις ε, χώρες. θέλουμε σωστές υπηρεσίες, τεχνικές επενδύσεις για την οικοδόμηση εσωτερικών και τοπικών δυνατοτήτων. Όμως η επένδυση στη, στη γεωργία οδηγεί σε μία σειρά από προκλήσεις από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται, για παράδειγμα, αν οι άνθρωποι ε, που, ε, που, που, που εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη γη, εκτοπίζονται και υφίσταται έξωση χωρί να του στηθεί η γνώμη του, χωρί να έχουν εναλλακτική λύση και χωρί ε, αποζημίωση. Επίση, παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα εάν τα τοπικά εισοδήματα δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την, τη μείωση του εισοδήματο λόγω της, της αύξησης των εισαγωγών, για παράδειγμα. και, λόγω του γεγονότο, για παράδειγμα, ότι έρχονται στην αγορά φθηνότερα προϊόντα, τα οποία οποία ε, παράγονται ε, αλλού σε ε, πιο ανταγωνιστικές και πιο εκτατικές. Επίσης το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, όταν παραβιάζει το δικαίωμα αυτό, όταν παραβιάζει το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή, σε τοπικό επίπεδο το δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά, το δικαίωμα της ενημέρωσης και της πληροφόρησης. So what obligations όσον αφορά τις υποχρεώσεις των κρατών και θα χρησιμοποιήσω το δικαίωμα στο φαγητό, ε, στην τροφή, σαν ένα ε, παράδειγμα. Αυτό το δικαίωμα αναγνωρίζεται σε διάφορα μέσα. Ε, και συνολικά στο Διεθνές Σύμφωνο για, οικονομικά, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Στο Γενικό Σχόλιο 11 της Επιτροπής για τα Οικονομικά, Κοινωνικά ε, και Πολιτιστικά Δικαιώματα. Όλοι θα πρέπει να φροντίζουν για την πρόσβαση ε, στο βασικό δικαίωμα στο φαγητό, ε, που είναι σε επαρκή ποσότητα και, στην κατάλληλη ποιότητα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πείνα των ανθρώπων. Το κράτος υποχρεούται να μην παραβιάζει την δυνατότητα των ατόμων και των ομάδων ε, να έχουν πρόσβαση στην τροφή. Αυτή είναι μια υποχρέωση που θα πρέπει να τηρεί το κράτο. Επίσης, θα πρέπει να παρεμποδίζει άλλου και ιδιαίτερα ε, σε ιδιωτικό επίπεδο όσον αφορά τι εταιρείε, για παράδειγμα, ε, που ε, προσπαθούν να στερήσουν από τα άτομα το δικαίωμα αυτό. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύεται με ενεργητικό τρόπο η δυνατότητα των ανθρώπων να μπορούν να θρέψουν τον εαυτό τους. Επίσης υπάρχουν υποχρεώσεις σε επίπεδο λήψης απόφασης και διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα, μη διακριτική μεταχείριση, επαρκής πρόοδος, συμμετοχή και σωστές δράσεις αποκατάστασης. So what could be done τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να έχουμε μια πιο υπεύθυνη, υπεύθυνη επενδύσεις στη γεωργία. Πρώτα απ' όλα πιστεύω, και αυτό αναφέρθηκε και από ε, τον προηγούμενο μιλητή, πρέπει να προωθήσουμε την προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επενδύσεις στη γεωργία. Και εδώ συμπεριλαμβάνουμε φυσικά και τις επενδύσεις στους φυσικούς πόρους. Ε, αυτό σημαίνει τουλάχιστον το σεβασμό των 11 αρχών ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, που, που αναφέρθηκαν από τον ε, ειδικό, ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στο φαγητό και οι 7 αρχές για τις υπεύθυνε επενδύσεις στη γεωργία. Ε, που έχουν αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει επίση ότι θα πρέπει να καθοριστούν υποχρεωτικέ λειτουργικέ κατευθυντήριε γραμμέ ε, και μοντέλα ε, και συμβάσει πρότυπα για τι επενδύσει στη γεωργία και οποιαδήποτε χρηματοδότηση, ιδιαίτερα από το δημόσιο, να συνδέεται με το σεβασμό αυτών των αρχών που υπάρχουν τώρα και είναι διαθέσιμες. Επίσης, προστασία των νομικών δικαιωμάτων των φτωχών, συμπεριλαμβάνοντας και την ε, πρόσβαση σε σωστού μηχανισμού επανόρθωση εάν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Επίση, πρέπει να δούμε τα ευρύτερα ζητήματα τα οποία ε, επιδρούν ε, στις ξένες επενδύσεις στη γεωργία. Δηλαδή, οι επενδύσει θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις εθνικέ στρατηγικές ανάπτυξη. και ο ειδικό εισηγητής για το δικαίωμα στην τροφή ζητά μια στρατηγική για την υλοποίηση του δικαιώματο στο φαγητό. Ε, αύξηση εισοδημάτων. Μια στρατηγική που να αυξάνει τα εισοδήματα και να μην οδηγεί σε μεγάλη παραγωγικότητα. Επίση, τα ευρύτερα ζητήματα τα οποία αφορούν τη διερεύνηση ε, συστημάτων παροχή κινήτρων για επιχειρηματικά μοντέλα συγκεκριμένα τα οποία συνδέουν ε, την επιχείρηση με του παραγωγού. Ε, για βιώσιμη ε, προμήθεια ε, αλλά και βιώσιμα εισοδήματα στους γεωργούς χωρίς μεταφορά των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας. Τέλος, ρύθμιση των παγκόσμιων αγορών για, ως προς τα αγροτικά προϊόντα και το εμπόριο των τροφίμων. Και εδώ θα μπορούσε να φερθεί το παράδειγμα των επιδοτήσεων. Μια διαδικασία αυτή θα, θα, θα οδηγήσει σε ένα πιο υπεύθυνο εμπορικό καθεστώς καθεστώς εμπορίου. Τέλο, θα πρέπει να γίνονται αξιολογήσεις αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά τι επενδύσεις αυτές για την εξασφάλιση του σωστού επιμερισμού των ε, κερδών. Και αυτό πρέπει να γίνεται πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά ε, ε, την ολοκλήρωση των επενδύσεων στη Γεωργία. Για όσοι ενδιαφέρεστε ε, στην, ε, ε στην, εμβα... περαιτέρω εμβάθυνση του ζητήματο, πέραν όλων αυτών των δημοσιεύσεων που αναφέρθηκαν μέχρι στιγμή και που θα αναφερθούν και από του επόμενου ομιλητέ, προετοίμασα ένα μικρό κατάλογο βιβλιογραφία που μπορεί να σα δώσει τελειώνοντα για να παραφράσω αυτό, τον, ε, τον συγγραφέα που ανέφερα και στην αρχή, σας αναφέρω ε, για την προστασία των ανθρώπων που ήδη βρίσκονται στο περιθώριο. Ε, δηλαδή, να μην δίνεται η δυνατότητα κερδοσκοπίας εκ μέρους των ξένων επενδυτών με τεχνητές αυξήσεις των τιμών ε, αυτό ε, έχει να κάνει με τα συγκρουόμενα συμφέροντα ε, όσον αφορά τη γη, ε, το, το είδωρ και, και την τροφή που οδηγούν σε τρομερές ε, καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπόριο ανθρώπων, πείνα κτλ. Τα ζητήματα αυτά είναι βασικά και το δικαίωμα στο φαγητό είναι βασικό. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό σήμερα και αν δεν φροντίσουμε την κοινωνική προστασία των ανθρώπων που έχουν δικαίωμα στη γη, στο νερό και στην τροφή, σίγουρα σπέρνουμε τους πόρους μελλοντικών συγκρούσεων και πολέμων. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία η παρουσίασή σας. Ο Μάικλ Τέριαν είναι ο επόμενος ομιλητής. Παρακαλώ, Μάικλ. Uh, uh, uh, Ξέρω όλοι έχουν κουραστεί. Εγώ άλλαξα τον τίτλο της παρουσίας μου την τελευταία στιγμή γιατί κάτι που είναι σημαντικό και εδώ και σε πολλές άλλες τέτοιες εκδηλώσεις ότι υπάρχει μια σύγχυση. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ της αρπαγής της γης, οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και την αγορά γη. Αυτά συχνά αλλοκαλύπτονται δυστυχώς σε ορισμένε περιπτώσει όχι. Θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να εξετάσουμε και τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ ανοίγω στη Διεθνή, ε, Συνδεσμό για τη Γη. Υπάρχουν εδώ τρει ε, οργανώσει, ορισμένε διακυβερνητικέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματο χάρη, ε, μεταξύ άλλων και άλλε οργανώσει, όπω οργανώσει των Ιωργών, ε, συνδικάτα, ε, οργανώσεις κοινωνία των πολιτών και ερευνητικά έργανα. Αυτό που μας ενώνει είναι μια κοινή ιδέα ότι η πρόσβαση και ο έλεγχο ε, της γης είναι ένα σημαντικό βήμα για να ξεπεράσουμε την ένδυα. Το πώς όμως είναι εκείνο που οδηγεί σε διαφορετικές απόψει στα μέλη μας. Οπωσδήποτε υπάρχει ενδιαφέρον στην επένδυση στη γη και αυτό έχει αυξήσει και το ενδιαφέρον στο όλο πρόβλημα που υπάρχει. έχουμε 35 οργανώσει εταίρου σε όλο τον κόσμο και μαζί τους προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Ε, είπαμε, ένας από τους επενδυτές μας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορισμένα από τα σημεία έχουν καλυφθεί. Θα δώσω ορισμένα στοιχεία μονάχα για το τι δεν πήγε καλά. Καταρχήν υπάρχει τεράστια έλλειψη διαφάνειας. Δεν γίνονται σε ανοιχτέ δια, ε, διαδικασίες, γίνονται στα παρασκήνια και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε ακριβώς ποιε είναι αυτές οι συναλλαγέ στον τομέα της γη. Ε, και υπάρχουν πολύ αντιφατικές ε, δηλώσεις, υπάρχουν αγροπολωσίες που δηλώνονται που δεν έχουν λάβει χώρα, άλλες όμως που γίνονται και δεν τις έχει μάθει ποτέ κανένας. Ένα άλλο επιστημονικό θέμα και κάτι που ενδιαφέρει την ε, Διεθνή Τράπεζα είναι η σχέση μεταξύ της, ε, του ενδιαφέροντος ε, των επενδυτών και της έλλειψης της διακυβέρνησης. Και υπάρχει εδώ μια αντίστροφη σχέση. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια τεράστια ε, πρόκληση ε, ότι οι επενδυτές πάνε εκεί όπου ξέρουν ότι θα έχουν τη λιγότερη νομική αντίσταση από εκείνους που ζουν επί τόπου. Γιατί είναι σημαντική η υγεία. Ο, πολλοί από εσάς ξέρουν, θα σας πω δύο-τρεις λόγους γιατί. Γιατί οπωσδήποτε είναι μια ε, πηγή στην οποία πάρα πάρα πολύ βασίζονται για, την, ε, για το καθημερινό τους είναι ένα βασικό ένα βασικό δικαίωμα ή μάλλον μια βασική ιδιοκτησία που έχουν για πολλούς χαρακτηρίζεται για την κληρονομιά είναι δηλαδή σημαντικό κοινωνικά ε, μάλιστα πολλές φορές η συμμετοχή κάποιων στην πολιτεία εξαρτάται από το κατά πόσον έχουν στα χέρια τους γη όχι και αν αλλάξει κανένα ε, τον τρόπο τον οποίο σχετίζονται οι πολίτες με τη γη, αλλάζουν πολλές φορές ε, ε, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η λειτουργία. Εγώ από την Ποτσβάνα είδα πω το θέμα τη γη ή μη γη, εξαρτήθηκε από το Απατχάιντ. Αλλά υπάρχει και το παράδειγμα της Φιλανδία που ακούσαμε. Ορισμένα σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να έχετε κατά νου κανένας με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους ποιος έχει πρόσβαση στη γη ή νόμιμο έλεγχο. 80% εκείνων που πεινούν στον κόσμο είναι σε αγροτικές περιοχές. Οι περισσότεροι δηλαδή που πεινάνε ζουν σε αγροτικές περιοχές. Το 70% όμως του, ε, των τροφίμων παράγοντα στον κόσμο παράγεται από μικρούς παραγωγούς. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος λοιπόν και τεράστιες ευκαιρίες. Γιατί είναι σημαντική αυτή η διαδικασία που έχει ενδιαφέρει και τα ΜΜΕ παγκοσμίω, γιατί καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι υγείας που συζητάνε δεν είναι κενές. Οι κενές είναι μέσα στην έρημο, στη Σαχάρα, στην Κόμπη. Εκεί δεν ενδιαφέρεται όμως κανένα να αγοράσει. Εδώ έχουμε παραγωγική υγιής που δεν έχει κάποιο στα χέρια του και που είναι η πιο φτηνή, η πιο φτωχοί, συγγνώμη, άνθρωποι του κόσμου. Πολλοί είπαν ότι πολλοί από του τομεί στου οποίου ενδιαφέρονται οι επενδυτέ ε, δεν υπάρχει αρκετή εναλλακτική δυνατότητα επιβίωσης, δεν υπάρχουν θέσεις απασχόληση και πολλοί προσπαθούν βέβαια να προσελκύσουν επενδυτέ στη χώρα του, ιδίω στην Ήπεθρο. Υπάρχουν δηλαδή και εκεί ευκαιρίες. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που γίνονται αυτή τη στιγμή και τα αρχικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι υπάρχουν ε, και κίνδυνοι πολύ μεγάλοι για ανητικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τεράστιοι κίνδυνοι, όπου πολλές φορές τα σχέδια αυτά μάλλον τις, τους κινδύνους, προς τους κινδύνους και όχι προς ευκαιρίες. Αυτό που θέλαμε να τονίσουμε είναι η χρήση της ε, κοινή ιδιοκτησίας, που εκτιμούμε ότι είναι μεταξύ ενός και δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων, είναι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτούς τους κοινούς, τις κοινέ γης. Συνήθως αυτό το εδάφιο ανήκουν στο κράτος. Αυτό πάλι σημαίνει ότι αυτά, αυτοί οι άνθρωποι είναι χρησικτήστες κατά κάποιον τρόπο. Είναι ο κύριος ο ε, κίνδυνος, η κύρια πηγή ανησυχίας. Γιατί από την άλλη μεριά οι χώρες αυτές όμως πουλάνε τις γης αυτές έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Δεν αναγνωρίζουν όμως το εθνικό δίκαιο των ανθρώπων που ζουν στη γη αυτή εδώ και πολλές πολλές γενιές. Θα πρέπει επίση να ξεχνάμε εκείνους τους πληθυσμούς που έχουν χρήση ε, κρατικής ε, χρήσης ε, της γης. Παραδείγματος χάρη η βοσκή. Αυτή είναι... Ε, εκείνοι που χρησιμοποιούν τεράστιες εκτάσεις και υπάρχει ο, ο αν τους αγνοήσουμε να καταστροφούν αυτές οι υγιές και επίσης το ίδιο ισχύει και για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Για να προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την ε, με αυτό το πίνακα. Vlog 739 so far, of which the majority are in Africa, 449, 182 in Asia, 12 in Eastern Europe. Έχουμε 409 στην Αφρική, 180 στην Ασία, 12 στην Ανατολική, 72 στην Λατινική Αμερική και 3 στην Οκεανία. Αυτά τα στοιχεία δεν σας τα δίνω έτσι για να σας πω ότι αυτές είναι οι μόνες ε, αγορές που έχουν γίνει. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω επιλέξει μια εταιρεία από την Ευρώπη για να δείτε ότι δεν είναι ο μύθος αυτό ότι οι Κινέζοι και λοιπά αγοράζουν δεν είναι σωστό. Έχουμε 50 επενδύσεις από εταιρείε που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από αυτέ 39 στην Αφρική, 3 στην Ασία, 7 στην Ανατολική Ευρώπη, 1 στην Λατινική Αμερική οι οποίε είναι για αγροκαύσιμα, 3 για αγροτικέ εκμεταλλεύσει, 4 για εξοπλίσει και 15 άλλε σε 27 χώρε. Και όπω σα είπα, αυτό είναι περίπου 700.000 εκτάρια ανά επένδυση. Πολύ σύντομο παράδειγμα όσον αφορά μήνε του επικοινωνίου. Έχουμε τη Μαζαβίκη εδώ που έχει από του πιο προοδευτικού ε, νόμου για τη γη στην Αφρική. είχαν επίσης μια πολύ επιθετική εξατία για να προσελκύσουν επενδυτές. Αριστερά βλέπετε το θέμα της ε, ε, αποδοτικότητας της γης. Τα πράσινα είναι τα πιο αποδοτικά προφανώς ε, τμήματα. Στα δεξιά, στο κίτρινο βλέπετε που υπάρχουν κοινωτικά δικαιώματα που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση. Το μπλε είναι επενδυτικά δικαιώματα που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση και βλέπετε ότι τελικά η, τα, τα δικαιώματα χρήση της γης έχουν δοθεί στις πιο ε, ξερές περιοχές. Αυτό δεν το ζητάνε όμως οι επενδυτές. Εκείνοι έχουν πάρει τα πράσινα τμήματα. Και τα κόκκινα που βλέπετε εδώ είναι οι χώρες, ε, τα τμήματα μάλλον στα οποία έχουν εργαστεί πάρα πολύ σκληρά βάσει του συστήματος Άθωνης που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν τα ίδια, οι ίδιες σχέσεις που έχουν δοθεί και στην κοινότητα και σε επενδυτέ. Αυτό δεν θα σας το παρουσιάσω. Είναι ένα παράδειγμα για την Τανζανία, το τι έγινε στην περίπτωση κάποιες συγκεκριμένες επενδύσεις. Θα τελειώσω την παρουσίασή μου με πέντε προτάσεις σαν αποτελέσματα της εργασίας μας που θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι ας πούμε να θέλουν να εμπλακούν. Καταρχήν θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν ξέρουμε αρκετά όσον αφορά το εύρος και τις ευκαιρίες και τους κινδύνους. Γιατί είναι σημαντική αυτή η έρευνα, γιατί παραδείγματος αναφερθήκαμε στην έλλειψη διαφάνειας. Εκτός αυτού, για φανταστείτε, εάν κάποιος ε, νοικιάσει μια γη για 99 χρόνια, αυτό μπορεί να αντιστραφεί αύριο. Πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια έρευνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα από την ΕΦΑΟ, Ευρώπα, ΦΙΑΝ, SNV και λοιπά. Μελέτες ε, από τη ΦΙΑ, παραδείγματος εκτός της Ευρώπα, για έξι χώρες στην Δυτική Αφρική, η SNV έχει αναλάβει πρωτοβουλίε έρευνα για 12 χώρε. Το κλαπ του Σαχέλ κάνει επίση κάποιε ενδιαφέρουσε ε, έρευνε στην Ασία και στην Αφρική και εμείς όπως σας είπα έχουμε 35 μελέτες που κάνουμε. Αυτό θα είναι η απαρχή της καλύτερης κατανόησης θα έλεγα. Χρειάζεται να καταλάβουμε πολύ καλύτερα και αν δούμε τις μεγαλύτερες έρευνες όπως αυτή από την ε, Διεθνή Τράπεζα, την ΦΑΟ και την ΙΦΑΞ που είναι πολύ ευρύς, θα πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα μελέτες από οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ε, πολίτες επιτόπου. Είναι πολύ καλό ότι η Ευρώπη μπορεί να εξετάσει από τη δική της πλευρά τι γίνεται, να υποβάλουν τα ερωτήματα που θέλουν και να δώσουν τις πληροφορίες τους στη συζήτηση. Οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει μια πιο επιφυλεκτική προσέγγιση, φαντάζομαι. Δεύτερον, θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί η καταγραφή των δικαιωμάτων καθεστώτος ιδιοκτησίας. Γιατί αν θα γνωριστούν αυτά τα δικαιώματα των τόπιων, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το αποτέλεσμα. Από αυτό κρίνεται ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει και δεν θέλουμε να χάσουν μόνο οι τόπιοι και θα χάσουν να χάσουν για πολλέ γενιέ. Αν αναγνωριστούν όμω τα δικαιώματά του στη γη θα μπορούν να κάνουν θεωρητικά τουλάχιστον μια ε, επιλογή αν θέλουν να δεχτούν την επένδυση ή όχι και αν τη δεχτούν κάτω από ποιου όρου. Τώρα πώ θα γίνει αυτό. Έχει ελεγχθεί ήδη πάρα πολύ καλά στο πρώτο πάνελ ότι είναι πολύ πιο εύκολο, φτηνότερο και πιο γλίγορο με τις τεχνολογίες που γραφτεί τα τελευταία χρόνια να γίνει η καταγραφή των δικαιωμάτων αυτών και τονίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωστούν και τα συλλογικά δικαιώματα. Εάν ορισμένες ε, κοινότητες που έχουν αναγνωσμένα συλλογικά ε, δικαιώματα θέλουν να αναγνωρίσουν και ατομικά δικαιώματα μπορούν να το κάνουν, αλλά καταρχήν θα πρέπει να προσπαστατεύσουμε τα δικαιώματα του συλλογικού, ε, της συλλογικής βάσης της ε, κοινότητας αυτής. Και οι κοινότητες θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι ε, επιμέρους ε, ιδιοκτήτες, οι ατομικοί ιδιοκτήτες. Αυτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Μάικλ για την παρουσίαση αυτή. Ο τελευταίο ομιλητή είναι ο Χένρι Σαραγκή, ε, γενικός συντονιστής της Λαβία Καπενσίνα. Uh, thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω πολύ και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε ως εκπρόσωπο του οργανισμού Λαβία Καμπεζίνα. Θα ήθελα εδώ πέρα να σας πω ότι εκπροσωπώ τους ακτήμονες, μικρούς καλλιεργητές, τους ε, φτωχούς αυτούς ανθρώπους που αναγκάζονται να επιβιώσουν μέσω των μοντέλων που αναπτύξατε, που παρουσιάσατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και ορισμένους από τους ομιλητές, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα σημαντικά σημεία, τα οποία θα ήθελα και εγώ να θίξω στην παρουσίασή μου. Για μένα η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική γιατί βρίσκομαι εδώ ενωπίων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Συγγνώμη, στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Στα πλαίσια του οργανισμού μου, Λαβία, Καμπεσίνα, προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να λύσουμε και εμείς το πρόβλημα. Πώς έχει ακριβώς το πρόβλημα. Ο αριθμός των ανθρώπων στον κόσμο που πεινάνε έχει αυξηθεί. Το 1996 είχαν, είχε δεσμευτεί η διεθνής κοινότητα για τη μείωση της πείνας. από τα 820 εκατομμύρια υποτίθεται ότι ο πληθυσμός αυτός θα μειωνόταν κατά το ίμιση. Αλλά έχουμε δει ότι έχουμε φτάσει πλέον το 1 δισεκατομμύριο ατόμων. Επίσης, στα πλαίσια των στόχων της χιλιετίας της των Ηνωμένων Εθνών είχε τεθεί ο στόχος της μείωσης της φτώχειας και βλέπουμε όμως ότι η ένδια έχει αυξηθεί αντί να έχει μειωθεί. Αν δούμε επίσης και το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Βλέπουμε πώς σε καθημερινή βάση τροποποιείται το κλίμα. Και βλέπουμε επίσης ότι έχουμε και το σημαντικό το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης. Εγώ προέρχομαι από την Ινδονησία όπου η οικονομική κρίση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και στο παρελθόν είχαμε μια οικονομική κρίση η οποία περιοριζόταν περισσότερο στην Ασία, ενώ τώρα βλέπουμε ότι η κρίση είναι παγκόσμια και έχει πλήξει και την Ευρώπη. Το πρόβλημα λοιπόν, οι ορισμένα τα προβλήματα που αναλύουμε δεν αφορούν πλέον μόνο κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και την ίδια την Ευρώπη και να επανέλθω στο σημαντικότερο ζήτημα για σήμερα. Εμείς ως μικροκαλλιεργητές, ακτήμονες μικροκαλλιεργητές, ασχολούμεθα εδώ και πάρα πολύ καιρό με το ζήτημα της αρπαγής της γης. Προέρχομαι, όπως σας είπα, από την Ινδονησία. Η Ινδονησία, όπως και πάρα πολλές άλλες χώρες που εκπροσωπούνται στην Λαβία Καμπεσίνα, πλήττεται ιδιαίτερα από την αρπαγή της γης. στο όνομα της εξαγωγής προϊόντων όπως ε, ο καπνός, το τσάι, το χαρτί. Υπάρχουν πάρα πολλά εκτάρια γης τα οποία αγοράστηκαν, αρπάχτηκαν θα έλεγα, από πολυεθνικές εταιρείες, από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα σφάλμα το οποίο μας έχει ε, κληροδοτήσει η απεικιοκρατία. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όμως το φαινόμενο της αρπαγής της γης. Ο φίλος μου από τη ΦΙΑΝ είπε πως ε, η απελευθέρωση ή η ιδιωτικοποίηση, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές για τη διαχείριση της γης έχουν συμβάλει στην αύξηση του φαινομένου της αρπαγής της γης. Από την οπτική γωνία της ε, Λανδία Καμπεζίνα βλέπουμε ότι πολλές φορές και οι πολιτικές της ίδιας της Παγκόσμιας Τράπεζας έχουν διευκολύνει την αρπαγή της γης από τις πολυεθνικές εταιρείε. Ένας από τους ομιλητές αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στους τίτλους ιδιοκτησίας. Μα οι τίτλοι ιδιοκτησίας τελικά ενισχύουν τους πιο ισχυρούς. Δίνουν τη δυνατότητα στις πολυεθνικές εταιρείε να αποκτούν τη γη και ουσιαστικά βάζουν σε υποδέστερη θέση τους μικροκαλλιεργητές. Στην Ινδονησία, στο Μεξικό και σε άλλες χώρες, ο τίτλος ιδιοκτησίας από τη στιγμή που θα εκδοθεί αυτόματα σημαίνει ότι η γη θα φύγει από τον μικροκαλλιεργητή και θα περάσει σε έναν πιο ισχυρό ή σε μία εταιρεία. Αναφερθήκαμε στην Μαδαγασκάρη, όπου αναφερθήκατε εσείς σε εκατοντάδες εκτάρια. Στην Ινδονησία βλέπουμε ανάλογα φαινόμενα όσον αφορά την αρπαγή της γης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, πολυεθνικές εταιρείες που αρπάσουν πλέον τη γη από τους καλλιεργητές. Στο παρελθόν, οι πολυεθνικές εταιρείες, αυτές που λειτουργούν διασυνοριακά και αυτές που άρπαζαν τη γη προέρχονταν από την Ευρώπη και από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Τώρα οι πολυεθνικέ εταιρείε έρχονται από την Κίνα, την Κορέα, ενδεχομένω και από την ίδια την Ινδονησία. ενδεχομένω και οι ίδιε οι Ινδονησιακέ εταιρείε να αρπάσουν αφρικανική γη. Γιατί υπάρχουν πλέον μεγάλε πολυεθνικέ εταιρείε που έχουν τη βάση του στην Ινδονησία και τη Μαλαισία και προσπαθούν να αποκτήσουν όλο και περισσότερη γη από την Αφρική. Υπάρχουν και αφρικανικές εταιρείες που, κάνουν, που ακολουθούν αντίστοιχες πρακτικές. Το πρόβλημα όμως είναι να δούμε πώς θα καταφέρουμε να επιλύσουμε το φαινόμενο αυτό, πώς θα καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε. Εμείς στα πλαίσια της Λαβία Καμπεσίνα έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να φύγουμε πλέον από το επικεκρατικό σύστημα διαχείρισης της γης και να περάσουμε σε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης και ιδιοκτησίας της γης. Βέβαια, δεν έχει επιτύχει το, το εγχείρημα αυτό σε πάρα πολλές χώρες. Έχουμε τα παραδείγματα της ε, Ιαπωνίας, του Βιετνάμ. Έχουμε και την Ευρώπη, όπου ορισμένες χώρες έχουν προχωρήσει με μια καλή γεωργική μεταρρύθμιση. Από το 1996 η Δία Καμπεσίνα στην Παγκόσμια Σύνοδο για τα Τρόφιμα είπαμε ότι προκειμένου να σώσουμε τον πλανήτη θα πρέπει να δώσουμε κυριαρχικά δικαιώματα στους μικροκαλλιεργητές. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου έχουμε πλέον καταστραφεί. Ο αριθμός των ανθρώπων που πεινάνε στον κόσμο όπως σας είπα, έχει αυξηθεί. Όχι επειδή έχει μειωθεί η παραγωγή τροφίμων, αλλά επειδή η παραγωγή τροφίμων βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στα χέρια των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Είναι οι μεγάλες βιομηχανίες που διαχειρίζονται πλέον την παραγωγή και τη διακίνηση τροφίμων παγκοσμίω. Στα πλαίσια της Λαβία Καμπεζίνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε προτείνει ένα συγκεκριμένο βιώσιμο μοντέλο οικολογικό για την ανάπτυξη της γεωργίας και για την ε, κατοχή της γης. Έχουμε δει ότι το μοντέλο το οποίο ακολουθείται στην Ασία δεν έχει στεφθεί με επιτυχία. Δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους γη. Θα θέλαμε λοιπόν να ακολουθηθούν οι σωστές πρακτικές στι άλλε υπήρου. Για παράδειγμα, στην Αφρική δεν θέλαμε να εξάγουμε στην Αφρική τι λαθασμένες πρακτικέ που έχουμε δει στην Ασία. Η Λαβία Καμπεζίνα λοιπόν ζητά μία μεταρρύθμιση της, των γεωργικών, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, όχι μόνο στην Ασία και στην Αφρική, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη. Ακούσαμε έναν Ευρωβουλευτή που είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε γη δεν έχουν δικαιώματα ιδιοκτησία. Πέρυσι, τον Δεκέμβριο, πήγα στην Κοπενχάγη, στη Σύνοδο για την Αλλαγή του Κλίματος. Η Δία Καμπεσίνα παρουσίασε εκεί πέρα την κατάσταση. Είπε πως σε καθημερινή βάση η γη φεύγει από τα χέρια των γεωργών, των μικροκαλλιεργητών. Φαινόμενο που βλέπουμε και στην Νότιο Κορέα και στην Ιαπωνία. Αλλά βλέπω ότι ακόμα και στην Ευρώπη σε καθημερινή βάση μειώνει το αριθμό των μικρών καλλιεργητών. Ελπίζουμε ότι και εσείς στην Ευρώπη θα υιοθετήσετε την δεύτερη γεωργική ε, μεταρρύθμιση και ότι θα φροντίσετε να αποφύγετε τις δεινές επιπτώσεις που, έχουμε, που σας περιέγραψα στην Ασία, που έχουμε βιώσει στην Ασία. Επίσης, ποια είναι η πολιτική η οποία ακολουθείται για τα βιοκαύσιμα, τα καύσιμα εκείνα τα οποία παράγονται από γεωργικά προϊόντα. Αν εσείς προωθήσετε την πολιτική που ακολουθείτε αυτή τη στιγμή για τα βιοκαύσιμα, τότε θα εξαφανιστούν τα δάση και από την Ασία και από την Ινδονησία πιο συγκεκριμένα και από τη Λατινική Αμερική. Γιατί παράγονται συγκεκριμένα προϊόντα μόνο και μόνο για να παραχθούν βιοκαύσιμα και όχι για να θρέψουν τους φτωχούς. Ελπίζω επίσης ότι η Επιτροπή αυτή αναφερόντας την κοινή γεωργική πολιτική στην Ευρώπη θα αναλογιστεί λίγο περισσότερο για το πώς θα μπορούσε να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική που θα προωθούσε περισσότερο την καλή διαβίωση των μικρών καλλιεργητών. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί περισσότερο με την παρακολούθηση των κλιματικών αλλαγών με την παρούσα κλιματική κρίση που έχουμε, έχουμε δει στην Ινδονησία ότι ε, στο όνομα της κλιματικής αλλαγής και της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής υπάρχουν προωθούνται πάρα πολλά αναπτυξιακά προγράμματα σε τρίτες χώρες όπως η Ινδονησία, όπως η Βραζιλία, όπου έχουμε ουσιαστικά αρπαγή γης. Έχουμε αρπαγή γης στο όνομα της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει επίσης να αξιολογήσετε τη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών εταιριών, των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη και να παρακολουθήσετε λίγο τη συμπεριφορά που έχουν εταιρείε αυτές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από το φίλο μου από την ΦΙΑΝ, να ζητήσει από τους αρμόδιους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνταχθούν περισσότερο με την πολιτική της ΦΑΟ προκειμένου να ακολουθήσουν και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συστάση που έχει κάνει η ΦΑΟ για την γεωργική μεταρρύθμιση και για την ιδιοκτησία της γης. Ορισμένες πολιτικές Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συντάσσονται με την πολιτική τη ΦΑΟ και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να προωθήσει την πρωτοβουλία της Βία Καμπεζίνα και να προωθήσει τα δικαιώματα των μικρών καλλιεργητών, των μικρών ε, χωρικών. Και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να προωθήσει κάποιες βέλτιστες πρακτικές που έχουν εντοπιστεί από τη δική μας οργάνωση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ Χένρι, σας ευχαριστώ όλους για τις τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Κοιτάξτε, 10 λεπτά έχουμε. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να πει κάτι. Έχετε το λόγο. Αν, δεν σας πειράζει να δίνω εγώ το λόγο, να δίνουμε εδώ το λόγο από το Προεδρείο. Ευχαριστώ. Ε, είπα πρώτα οι κυρίες γιατί δεν ήμουν και έτοιμος να πάρω το λόγο. Ε, και οπότε θα καθυστερήσω ένα λεπτό περισσότερο. Με εντυπωσίασε πολύ αυτά που ακούσαμε από την κυρία Ρούπανερ και τον κύριο Τέιλον νομίζω ότι πράγματι πρέπει να φύγουμε, να ξεφύγουμε τα ιδεολογικά πλαίσια. Ε, θυμάστε τι έλεγε ο την ιδεολογία. Ο καπιταλισμός είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο και ο κομμουνισμός είναι το αντίστροφο. Άρα λοιπόν, αν συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτή την πτυχή, δεν θα πάμε και πολύ, δεν θα προχωρήσουμε και πολύ μακριά. Θέλουμε λοιπόν μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Η δυσκολία που έχουμε είναι αυτό, αυτό που είπατε και συμφωνώ παρόλο που είμαι φιλελεύθερος, ε, συμφωνώ ότι στο γεωργικό τομέα δεν μπορούμε τα πάντα να τα επιλύσουμε με την αγορά. Υπάρχουν και δικαιώματα αλλά και συμφέροντα. Και το δικαίωμα στην διατροφή, παρόλο που δεν έχει τόσο κωδικοποιηθεί όσο τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά, αυτά που ε, δημιουργήθηκαν από τη Γαλλική Επανάσταση. μιλάω δηλαδή για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρώτη γενιά. Πάντω σίγουρα θα πρέπει ε, να διπλασιάσουμε τι προσπαθίε μα για να ορίσουμε τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Ε, από τα οποία αυτά τα δικαιώματα εξαρτάται και η επιβίωση τη πρώτη γενιά δικαιωμάτων σε αναπτυσσόμενε χώρε. Τη δυσκολία που έχουμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι οι θεσμικοί ε, πρωταγωνιστέ, τα κράτη, η Επιτροπή έχουν ω συνομιλητέ του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών. Και μόλις υπάρξει παραμικρή παρέκκληση από το πολιτικά ορθό, τα εμπόδια είναι ξεπέραστα. Το να πάει κανείς σε μια χώρα και να κάνει την επανάσταση σημαίνει ότι αν σε μια χώρα έχουμε μια επανάσταση, τότε χάνουμε πλέον ε, τους διάβλους επαφής, τις επικοινωνίες μας. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω, αλλά όσον αφορά αυτά τα οποία είπατε, για να σημειώσουμε πρόοδο, πρέπει να έχουμε κάποια σταθερά σημεία αναφοράς. Παράδειγμα, ε, ε, ε σας αναφέρω το παράδειγμα Πιζανή που αναφέρεται ε, ότι στο εξή, εάν θέλουμε να τρέφονται όλοι οι άνθρωποι, εάν θέλουμε σωθεί η ανθρωπότητα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη, τη γεωργία σε παγκόσμια κλίμακα. Το δικαίωμα στη διατροφή σίγουρα υπερτερεί και είναι υπεράνω των οικονομικών συμφερόντων, των επιμέρους οικονομικών συμφερόντων. Αν λοιπόν υπάρξει κατανόηση ε, όσον αφορά αυτή την πτυχή που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ρεαλιστική, τότε θα μπορούσαμε ίσως να σημειώσουμε πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή. Εάν δεν το πράξουμε, τότε ε, πραγματικά ε, όλα αυτά ε, έχουν να κάνουν ε, με, ε, θα, θα, θα ε, οδηγηθούμε σε άσχημες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα στη, στις αναφέρω τη Ζιμπάμπουε. δεν, δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. Ε, τώρα, σε ποιο βαθμό λοιπόν μπορούμε να είμαστε παρεμβατικοί και μεμβατικοί για να επιληθούν τα προβλήματα αυτά. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι στις ε, συμφωνίες εταιρική σχέσης με τις χώρες Αφρικής θα πρέπει να, να θίξουμε το πρόβλημα με τι κυβερνήσει. Γιατί νομίζω ότι σε τελευταία ανάλυση και οι ίδιε οι χώρε έχουν συμφέρον, οι αγρότες τους, που ε, είναι ε, το μισό του πληθυσμού τους, θα πρέπει να μπορούν να επιβιώσουν. Άρα πρέπει να το, να το θίξουμε το πρόβλημα αυτό. Πόσο θα κοστίσει? Πόσο θα κοστίσει? Πώς, πώς θα κόστιζε εάν αγοράζαμε τη γη για λογαριασμό αυτών που δεν έχουν τίποτα, αλλά που έχουν επάγγελμα, είναι, είναι αγρότες, είναι χωρικοί. Ποια θα, ποια ήταν η τιμή, το τίμημα όλων αυτών. Έχουμε, πρέπει να σκεφτούμε, έχουμε μια μελέτη του ΦΑΟ, τη συζητήσαμε πριν από λίγους μήνες. Εσείς αναφερθήκατε σε πολλές άλλες μελέτες, κυρίως ε, σε, ε, σε μία μελέτη ε, που έγινε από τις χώρες της Δυτικής Αφρικής και από, τον, και από την ομάδα... Το και από, την, και από το κλαμπ των Σεχελών και νομίζω ότι πράγματι είναι πάρα πολύ χρήσιμο λεφτά και θα έπρεπε να ακούσω την άποψη τη Επιτροπής όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Τι άποψη έχει και μέχρι πού μπορούμε να πάμε ε, ε, θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στο συγκεκριμένο τομέα ε, και να προστατεύουμε τη γεωργία. Άλλωστε, και στην ίδια την Ευρώπη. Έχουμε διαφορετικά κτηματολόγια και εγγραφή της ιδιοκτησίας στα διάφορα κράτη-μέλη ποικίλαν, όσα και τα κράτη-μέλη. Αλλά όλα αυτά προστατεύουν τους γεωργούς και ε, παρεκκλίνουν από την ελεύθερη πρόσβαση στην ιδιοκτησία. Δεν υπάρχει καμία χώρα. Κοιτάξτε, στη Γαλλία, για παράδειγμα, απαγορεύσαμε σε ορισμένε περιπτώσει ε, την αγορά γη από του αλλοδαπού, εκτό και αν ήταν εγκατεστημένοι ε, ω αγρότε στην γαλλική επικράτεια. Εάν δεν, μέχρι πρόσφατα, εάν δεν πληρούσαν τον όρο αυτό, ακόμα και σήμερα νομίζω μερικέ περιπτώσει, δεν είχαν δικαίωμα πρόσβαση και αγορά γη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δεσμευτούμε προς, τα, προς την κατεύθυνση αυτών των σημείων που και, που και αναφέρετε, τότε πραγματικά ε, δεν, τουλάχιστον στην Ευρώπη δεν θα, ξεφ, ε, ξεφεύγαμε και πολλά πράγματα που ήδη έχουν γίνει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφη έχει το λόγο. Ευχαριστώ ε, για, τα, για αυτά τα οποία είπατε. Εγώ έχω μια ε, ρεαλιστική ερώτηση. Σύμφωνα με την άποψή σας και απευθύνουμε σε όλους τους ομιλητές. Ε, πέραν τη μεταρρύθμιση κοινή αγροτική πολιτική. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που είπατε. Αλλά ποια εργαλεία θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ε, ε, ότι, ότι, ότι η χρησιμοποίηση τη γη θα γίνεται ει βάρο των πλέον αδυνάμων και των πλέον φτωχών. η αξιοποίηση τη γη. Πώ θα μπορούσαμε εμεί να σημειώσουμε πρόοδο στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσουμε αυτό το σφετερισμό, αυτή την απαρπαγή τη γη. Ευχαριστούμε. Άλλες ερωτήσεις. Να κάνω κι εγώ κάποια ερώτηση. Ναι, πρώτα η συνάδελφος να κάνει την ερώτησή τη. Ε, θα ήθελα να σας κάνω, ε, ε, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, θα ήθελα να πω και είναι πολύ καλό το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η έκθεση ε, για να έχουμε πιο συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία αναχώρε. Γιατί εγώ πρόσφατα εργάστηκα με την κυβέρνηση τη Μοζαμπίκη στο γεωργικό τομέα και εξετάσαμε τα βιοκαύσιμα, τα δάση, τα διάφορα προγράμματα στον τομέα των τροφίμων και μα εξέπληξε ιδιαίτερα τα αριθμητικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι 5 ως 8 εκατομμύρια εκτάρια έδωσε ε, η κυβέρνηση της Μοζαβίκης ε, σε, σε διάφορα συμφέροντα. Ενώ 50.000 ήταν αυτά που δόθηκαν στον κόσμο. Καταλαβαίνετε τα, τα, στοιχεία είναι πολύ ε, σημαντικά. Δεύτερον, η συζήτηση αυτή για την αρπαγή της γης συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με τι ανεύθυνε κυβερνήσει. Δεν είναι αυτή η εμπειρία μου. Ε, εντάξει, έχω στο μυαλό μου ιδιαίτερα τη Μοζαμπίκη. Δεν ξέρω τι έγινε με την Καμπότζη. Αλλά υπήρξαν σοβαρέ ανησυχίε σε επίπεδο κυβέρνηση ε, όσον αφορά τη χώρα αυτή. Σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, στο Συμβούλιο των Υπουργών. Ε, είπαν πώ θα κοιτάξουμε τα εγγόνια μα ε, ε, κατά πρόσωπα και θα του πούμε ότι ε, στον αγώνα τη απελευθέρωση αγωνιστήκαμε ιδιαίτερα για να απελευθερωθεί η χώρα μα και τελικά την εκχωρήσαμε στου ξένου. Άρα απαιτείται περισσότερο διάλογο και με τι ίδιε κυβερνήσει. Γιατί ε, ε, όσον αφορά τι παρουσιάσει, εγώ δεν άκουσα ε, να αναφέρεται τίποτα στην άποψη των κυβερνήσεων. Δηλαδή, προποθέτουμε ότι οι κυβερνήσει απλά χαρίζουν τη γη, ε, εκχωρούν τη γη του. Και βεβαίω, εγώ αναφέρομαι στη Μοζαμβίκη για άλλη μια φορά. Και ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα μπορούσε να εξετάσει τι μπορεί να κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σκεφτούμε εδώ τη συνέπεια τη προσέγγιση ανάμεσα στι διάφορε γενικέ διευθύνσει τη Επιτροπή. Γιατί ε, όσον αφορά και κάποιες άλλες, στους άλλους οργανισμούς ανάπτυξης. Να πω ότι υπήρξε ασυνέπεια ανάμεσα στα διάφορα τμήματα. Ένα τμήμα προωθούσε την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα ε, και την άρση των γραφειοκρατικών ε, και διοικητικών εμποδίων για τη διευκόλυνση των επενδύσεων ε, και την απομάκρυνση από τον κυβερνητικό έλεγχο και, από την, και σε μια άλλη υπηρεσία προωθείται το αντίθετο. Δηλαδή ότι πρέπει να είναι το κράτος πιο αυστηρό και να προσπαθεί να επιλέγει τις καλές επενδύσεις. Άρα νομίζω ότι και οι ίδιες, και οργανώσεις πρέπει να είναι συνεπής με το ίδιο τον Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς. Ε, θέλω και εγώ να κάνω μία ερώτηση και θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε μέχρι τις 6 και 10. Κύριε Τέιλορ, ε, δεν ακούσαμε καθόλου τη λέξη διαφθορά, ενώ ακούσαμε στοιχεία. Πώς το κράτος δίνει χρήματα στον ιδιωτικό τομέα και ξεπερνά ε, τις δικές τους δικούς του νόμους. Ε, επίσης, ε, ε, ε, νομοθεσία για τα ανθρωπιστικά δικαιώματα με βάση τη γη. Στο δικό μου σύνταγμα αναφέρεται το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, κατοχυρώνοντας δικαίωμα. Ίσως θα μπορούσαν και κάποιοι άλλοι ομιλητέ να πούν λίγο περισσότερο για το ζήτημα αυτό. Γιατί όταν μιλάμε για την αναθεώρηση του μέσου αναπτυξιακή συνεργασία, που είναι βασική νομοθεσία για την αναπτυξιακή ε, βοήθεια, δεν πρέπει να δούμε και αυτή την πτυχή και με ένα κάποιο διαφορετικό, κάπως διαφορετικό τρόπο. Και ο Μάικλ επίση αναφέρθηκε ε, η εξέταση ε, του αντικτύπου των διαφόρων δυνατοτήτων. Ποιο θα κάνει την έρευνα αυτή. Έκανε κάποια έρευνα προ την κατεύθυνση αυτή η Επιτροπή. Αναφέρατε ορισμένε οργανώσει που έχουν ε, ασχοληθεί με, τέτοιες, με τέτοιο ερευνητικό έργο. Ε, λοιπόν, να σα δώσω το λόγο, κύριε Ντίβα, για δύο λεπτά και μετά θα δώσουμε το λόγο στο Μίλτερ. Ο Μάικλ είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο τετραγωνίζει τον κύκλο από πολιτική άποψη. Με την έννοια ότι, θα κάνουμε, μια, ότι κάνουμε εδώ μια πολιτική συζήτηση. Ο Μάικλ ε, στηρίχθηκε στην υπόθεση ότι οι κυβερνήσει έχουν ε, το απόλυτο νομικό δικαίωμα να δίνουν μεγάλα τμήματα γης σε ξένους. Και να στερούν από την ιδιοκτησία του δικού τους πολίτες. Επειδή δεν καταχωρήθηκαν ως ιδιοκτήτες οι πολίτες τους. Και ο μόνο τρόπο τον οποίο μπορώ να σκεφτώ ε, ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να σταματήσουμε ε, τι κυβερνήσει από το να δίνουν αυτά τα μεγάλα ε, τεμάχια και όταν τα δίνουν αυτά τα μεγάλα κομμάτια γη. Ε, τότε κοιτάξτε, ε, αυτό συμβαίνει. Άρα λοιπόν, εάν οι κυβερνήσει στερούν την ιδιοκτησία από το λαό τους και δίνουν αυτά τα αυτές οι ιδιοκτησίε νόμιμα στους, στους άλλους και δεν προβλέπεται τίποτα από την νομοθεσία, ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε αυτή την πρακτική είναι να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα αυτό και να απαιτούμε όλοι όσοι ζουν στη συγκεκριμένη περιοχή, σε κοινότητες, σε ομάδες ή σε ατομική βάση, να εγγραφούν, να καταχωρηθούν ως ιδιοκτήτες συγκεκριμένη γης. Ωραία. Ποιο μέλος ε, του πάνελ θέλει να απαντήσει. Ξεκινάμε. Ένας-ένας από τα ε, δεξιά. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο όσον αφορά το ερώτημά σα, για συγκεκριμένα ε, βήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη σα μίλησα για αυτή τη διαδικασία των εθελοντικών κατευθυντηρίων γραμμών. Ναι, εθελοντικέ, το καταλαβαίνω, στη ΦΑΟ. Αλλά ένα από του σκοπού ε, και ο σκοπό του Ολιβιέ Σούτερ του ειδικού ε, εισηγητή για το δικαίωμα στο φαγητό, στα τρόφιμα, είναι όλες οι υποχρεώσει στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με το ζήτημα της γη να συγκεντρωθούν και να χρησιμοποιηθούν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ε, ως μέσον, ε, να χρησιμοποιηθούν συνολικά και στα πλαίσια της αρπαγής της γης. Ίσως αναφορά το τελευταίο σημείο, και το πρόβλημα της, ε, της, ε, της έλλειψης δικαιώματος όταν δεν έχουν εγγραφεί και καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτες. Υπάρχουν παραδείγματα όπου έχουν καταχωρηθεί οι άνθρωποι αυτοί, αλλά είδαμε στην Καμπότζη ότι δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι η τυπική πλευρά. Ακόμα και αν έχουν εγγραφεί ε, τα δικαιώματα αυτά, και εδώ φτάνουμε στη διαφθορά, η κυβέρνηση, στη διαφθορά και σε άλλα συναφή ζητήματα, παρόλα αυτά, παρά το γεγονό ότι υπάρχουν ε, ε, τα χαρτιά κτλ., δίνει τη γη αυτή η κυβέρνηση. Δεν είναι λοιπόν πανάκια η καταχώρηση. Και να, θεωρούμε, να θεωρούμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο βρήκαμε τη λύση. Ευχαριστώ. Θέλετε να πείτε δύο λόγια, Χένρι, εν είδη I think uh, to solving this issue. Κοιτάξτε, σαν αυτό το ζήτημα αυτό, δεν μπορούμε να το βλέπουμε μόνο από την νομική σκοπιά. Πρέπει να δούμε και το γιατί ε, έγινε αυτή η αρπαγή της γης. Γιατί η κυβέρνηση δίνει στους ξένους τη γη. Γιατί ο τίτλος δεν σημαίνει ότι αυτόματα έχουν και την εγγύηση οι άνθρωποι αυτοί. Το έχω δει εγώ σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί ορισμένε πολυεθνικές δεν αρπάζουν μόνο τη γη. Γιατί πληρώνουν γι' αυτό. Δίνουν ένα αντίτιμο. Αποζημίωση. Και με το χαρτί ε, γίνεται και πιο εύκολα η αγοραπολισία. Άρα, να μην προσεγγίζουμε το ζήτημα μόνο από την νομική σκοπιά, να εξετάζουμε και περισσότερο ε, την ευρύτερη εικόνα, τη συνολική εικόνα της κατάστασης. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Um, following my previous... Κατάβουν αυτό που ερωτήθηκαν ποια είναι τα συγκεκριμένα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Θέλω να πω ότι και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στον διεθνή αυτό διάλογο που θα οδηγήσει σε κάποιε εθελοντικέ καθεσβήνες γραμμέ. Αυτό είναι βέβαια μία πλευρά τη εικόνα. Υπάρχουν και τεράστιες δυνατότητες επενδυτών Υπάρχουν όμως και μετά κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν εάν δεν ακολουθούν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές. Θα πρέπει λοιπόν να τις καταστήσουμε λειτουργία κατά το δυνατόν και επίσης θα πρέπει να σχετίσουμε την δημόσια χρηματοδότηση για τις επενδύσεις στην ε, αγροτική γη στην χρήση και εφαρμογή αυτών των αρχών. Ένας συγκεκριμένο τρόπος είναι είμαστε σίγουροι ότι οι διεθνείς υπηρεσίες ε, ανάπτυξης, όπως οι η Διεθνή Τράπεζα και άλλες ε, οργανώσεις, εφαρμόζουν τις κατευθύνσει γραμμέ επίσης στις συναλλαγές του ε, στη Γεωργία, πράγμα που δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. για να καταστεί το θέμα πιο λειτουργικό. Βέβαια, εσείς ως βουλευτές είναι σημαντικό να ζητάτε λογοδοσία του εκτελεστικού ε, οργάνου. Και πραγματικά είναι καλό να υπάρχουν αυτές τις, αυτά τα benchmarks. Ε, όσον αφορά το θέμα ότι οι κυβερνήσεις ε, δρούν νόμιμα όταν χαρίζουν αυτές τις γιές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περισσότεροι έχουν αναλάβει την υποχρεώση να τηρήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και έτσι θα μπορούν να το ζητηθούν και ε, λόγοι να απαντήσουν. Ο Μάικλ, συγκεκριμένα μέσα στο τέλος παρουσίας μου ανέφερα δύο. Οι άλλοι τρει που θα ανέφερα ήταν ε, η υποστήριξη των κυβερνήσεων στην Νότη να, κάνουν ε, καλύτερες να πάρουν καλύτερες αποφάσεις γιατί, ας πούμε, παραδείγματο, χάρη, ναι, δεν υπάρχει καμία εγγύηση αυτή τη στιγμή ούτε για την ε, εξαγωγή τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, Εκτό από τις ορισμένες επιπτώσεις. Είναι αλλιώς πραγματικά είναι αληθές ότι πολλές φορές ε, ορισμένες κυβερνήσεις είναι απεγνωσμένες για να υπάρχει ανάπτυξη. Δεν έχουμε τα μέσα για να πετύχουμε μια καλή, ε, μια καλή συμφωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι αποφάσεις για τη γη να λαμβάνονται με όλους τους ενδιαφερόμενους. Ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην κοινωνία των πολιτών στις χώρες αυτές να είναι τμήμα της απόφασης. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει πολλές από αυτές τις οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, πράγμα που είναι πολύ καλό. Είναι σημαντικό να υπάρχει επιτήρηση από τις κοινωνίες των πολιτών. Είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ καλό, σε ορισμένες περιπτώσεις όμως όταν γίνεται πνευματική αρπαγή της γης, οι χώρε αυτέ δεν σέβουν καν τον, το ίδιο το Σύνταγμα. Πώ μπορούμε να περιμένουμε να σεβαστούν διεθνεί συμφωνίε. Μόνο με την ενδυνάμωση τη κοινωνία των πολιτών στι χώρε αυτέ θα μπορούμε να αποφύγουμε τι αρνητικέ αυτέ επιπτώσει. Εκτό αυτού, τελευταίο σημείο χρειάζεται η, μια διεύρυνση του διαλόγου. Αυτή τη στιγμή έχουμε το διάλογο στα πλαίσια του Α, υπάρχει όμως η UNCTAD και τη Διεθνής Τράπεζα με μια σειρά προτάσεων που και αρχών που προτείνουν για την πρόθεση αυτών. Και έχουμε επίση τη Βία Καμπεσίνα που λέει από την άλλη μεριά ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές αρχές γιατί αυτό υποσκάπτει ίσως την, τα τοπικά ε, συστήματα παραγωγής. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει πιο ε, αναλυτικά και σε ευρύτερη βάση. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ το θέμα της, ε, ε, των δικαιωμάτων ιδιοκτησία, καθώ η ιδιοκτησία και την αρπαγή τη γη έχει αναγνωστεί σαν πάρα πολύ σημαντικό σε μια πρόσφατη ε, ανακοίνωση που είχαμε εκδώσει. Εκεί είχαμε αναφέρει επίσης την υποστήριξη μας για την εργασία πάνω σε κατευθύνες γραμμές που πρέπει να αναπτυχθούν. Και υποστηρίζουμε επίσης την εφαρμογή σε όποιες χώρες είναι δυνατόν των αρχών της, του δικαιώματος σε τροφή. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι κατά τη γνώμη μας το θέμα της διαφάνειας. Η διαφάνεια μπορεί να υποστηριχθεί και από εκεί μας σκοπιά και ο Μάικαλ το ανέφερα. Ο παρέμβαση χάρη με την υποστηρίξη τη κοινωνία των πολιτών και άλλων οργανώσεων, όπω οργανώσεων των παραγωγών, των αγροτών, που μπορούν να προωθήσουν τα δικαιώματα αυτά των αγροτών και τη χρήση της γης. Με έρευνα συγκατάσταση και πιο ουσιαστικά στοιχεία ή με την υποστήριξη της ε, καταγραφής ε, των ε, δικαιωμάτων στη γη κλπ. Πολλά μπορούν να γίνουν λοιπόν. Σημείωσα επίσης το θέμα της συνοχής ε, της πολιτικής και θα το λάβουμε υπόψη μας σε σχέση με άλλες υπηρεσίες ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις εν λόγω γενικές διευθύνσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, και πρέπει να έχετε κατά νου το θέμα για την ευρύτερη διαβούλευση. Πού το εννοείται αυτό? Αυτή τη δημοκρατική διαδικασία που το εννοειται αυτο αυτη η δημοκρατικη διαδικασια που μπορουμε να φανταστούμε, ούτως ώστε να εμπλακούν πραγματικά οι πολίτες όλοι. Ναι, ναι, ναι, ναι, φυσικά. Μα φυσικά. Πάρα πολύ ευρύ διάλογο είναι πάντα πάρα πολύ καλό. Άρα σα ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ μακρύ απόγευμα, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Με δύο πτυχέ ε, του θέματο και ήταν νομίζω μια πολύ χρήσιμη ακρόση. Θα ήθελα να ευχαριστώ όλου του που ήταν στα πάνελ, του συναδέλφου που συνέβαλαν. Ξέρω ότι υπάρχουν ταυτόχρονα πάρα πολλέ συνεδριάσει, ορισμένοι πηγαίνουν έρχονται λοιπόν και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του βοηθού, την Κομισιόν βέβαια. Σα ευχαριστούμε ιδιαίτερα και ευχαριστώ και του διερμηνεί και όλοι όσοι προετοίμασαν συνεδρία στη Γραμματεία ιδιαίτερα. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εδώ ολοκληρώνουμε τη συνεδρία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω ευχαριστώ. and good night from him.